Καλησπέρα σας συνάδελφοι. Ας αρχίσουμε παρακαλώ τη συνεδρίασή μας γιατί είναι αρκετά πιεσμένο το πρόγραμμά μας και είναι μεγάλες οι προσδοκίες. Ακούγεται Έχουμε υψηλές προσδοκίες από τον διαρθρωμένο διάλογο με τον Επίτροπο. Φάνηκε και από την πληθώρα ερωτήσεων που στείλαμε και αυτό το κάναμε για να είναι καλά προετοιμασμένος ε, ο Επίτροπος και να μπορέσει να απαντήσει. Ε, βέβαια, έχουμε πολλά και διάφορα προβλήματα. Θα είναι δύσκολο να τα καλύψουμε όλα σήμερα. Ναι. Ε, πριν όμως περάσουμε στο διαρθρωμένο διάλογο θα ακούσουμε την παρουσίαση από τον Επίτροπο για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Πρώτα όμως να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη, να πούμε ότι έχουμε σε 18 γλώσσες διερμηνία, έγκριση των πρακτικό 13 Μαρτίου, 20 και 21 Μαρτίου με την συνηθισμένη διαδικασία ως προς τις ανακοινώσεις αυτά. Και να περάσουμε στην παρουσίαση από τον Επίτροπο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Να καλωσορίσω καταρχήν τον Επίτροπό μας. Όπως είπα, κυρίως θέμα της σας διάταξη είναι ο διαρθρωμένος διάλογος, γιατί ήδη συναντήσαμε για, στα πλαίσια του διαρθρωμένου διαλόγου τον Επίτροπο Βιτένης Αντριουκάητης και σήμερα πριν περάσουμε στο διαρθρωμένο διάλογο, θα ακούσουμε την παρουσίαση από τον Επίτροπο Χόγκαν της πρότασης για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Αυτό και θα δώσω μέσω στο λόγο στον Επίτροπο για την παρουσίαση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, αξιότιμα μέλη. Είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας κάνω μια σύντομη παρουσίαση για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης που εγκαινιάστηκε σε 7 Δεκεμβρίου του 2016 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήδη έκανα τη σχετική παρουσίαση στο Γεωργικό Συμβούλιο και πολλοί συνάδελφοι έκαναν αντίστοιχες παρουσιάσεις σε άλλες ε, κοινοβουλευτικές επιτροπές. Πριν σας κάνω μια σύντομη παρουσίαση με PowerPoint, που σας την έχω στείλει κιόλα, θα ήθελα να κάνω κάποια εισαγωγικά σχόλια για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης δίνει ευκαιρία για εθελοντισμό στους νέους για να κάνουν μαθητείες και ασκήσεις σε πολλούς τομείς και να δείξουν την αλληλεγγύη τους. Τέτοιες ε, δραστηριότητε αλληλεγγύης μπορούν να γίνουν σε πολλούς και διάφορους τομείς, όπως τη γεωργία, την αγροτική ανάπτυξη, την περιβαλλοντική προστασία, ε, αποτροπή θεομηνιών, όπως είναι ανοβρία, πυρκαγιές δασών, πλημμύρες, ε, ε, θέματα διατροφής, ε, παιδείας, ε, υγείας, ένταξης των προσφύγων ή εδαφικής συνοχής. Συνεχίζεται αυτή η πιλωτική φάση και θα ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2017 και μάλιστα 1,8 εκατομμύρια είναι η συνδρομή μας στα πλαίσια της περιβαλλοντικής προστασίας της, της ζώνης του Natura 2000. Συνεχίζεται τώρα ε, η πρώτη φάση. Στι αρχέ του επόμενου έτου θα πρέπει να ξεκινήσει η δεύτερη φάση. Και μάλιστα η σχετική πρόταση θα υιοθετηθεί στι 24 Μαου από, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για αυτή τη δεύτερη φάση έχει προβλεφθεί ε, η ΚΑΠ να συμβάλλει με το ίδιο ποσό όπως και στην πρώτη φάση. Η συμβολή αυτή ε, του 1,8 δις Στη φάση, στη φάση αυτή θα συμβάλλει στην κάλυψη των ευρύτερων αναγκών της Ευρωπαϊκής Κοινωνίας και στην, την υλοποίηση των στόχων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θέλουμε ε, να φέρουμε πολλούς νέους κοντά στη γεωργία, την αγροτική ανάπτυξη, το περιβάλλον και την τασοκομεία. Και φυσικά δεν πρέπει να περιοριζόμαστε μόνο σε κεντρικά, ε, σε κεντρικά διαχειριζόμενες δράσεις. Θέλουμε επίσης ε, σε άλλους τομείς που χρηματοδοτούνται από την κυνηγιορική πολιτική να αναπτυχθούν ε, δραστηριότητες εθελοντισμού. Και μάλιστα ήδη ε, εκτελούνται και ε, δρομολογούνται πολλά προγράμματα στα πλαίσια της αλληλεγγύης, όπως είναι η ένταξη και υποδοχή προσφύγων, αποφυγή θεομηνιών, φυσικών καταστροφών και μάλιστα γίνεται έμπρακτη εφαρμογή των δραστηριοτήτων αυτών του, Σώματο αλληλεγγύη στην, στην Ήπεθρο. Έχουμε και θέματα όπω ε, τεχνική αρρωγή, ε, κατάρτιση και ε, στελέχωση του, του σώματος ώστε να επιτελεί συγκεκριμένα καθήκοντα. Και βέβαια εξαρτάται από τα κράτη-μέλη πώς θα αξιοποιήσουν τις δραστηριότητες, που τους τις ευκαιρίες που τους δίνει αυτό το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Θέλω λοιπόν, αν το επιθυμείτε και φυσικά και εσείς, να προωθήσετε αυτή την πρωτοβουλία, γιατί θεωρώ ότι το Σώμα Αλληλεγγύης θα ενισχύσει την αλληλεγγύη και την κατανόηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο κρατών μελών. Και να περάσουμε στην παρουσίαση με το PowerPoint για να σας δώσω περισσότερες πληροφορίες και το γενικό υπόβαθρο αυτού του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Όπω είπα, στόχο τη παρουσίαση είναι να κάνω γνωστό αυτό το πρόγραμμα, αυτή την πρωτοβουλία που βρίσκεται ακόμη σε πιλωτική φάση με στόχο να εμπλέξει 100.000 νέους ε, και να ενταχθούν σε αυτό το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης μέχρι το 2020 για να αποκτήσουν πείρα, να αναπτύξουν δεξιότητες και να συμβάλλουν στην κοινωνία. Περίπου 29.000 έχουν ήδη εγγραφεί στο σώμα αυτό και προσπαθούμε να κάνουμε μια αντιστοίχηση μεταξύ των εθελοντών και των διαφόρων φορέων. Ο πρώτος ε, ε, Γάλλος εθελοντής πήγε στην Ουγγαρία και δύο μαθητευόμενοι, Πορτογάλος και Ιταλός, έχουν ήδη τοποθετηθεί στο Βέλγιο. Και μάλιστα μετά την υιοθέτηση της σχετικής νομοθεσίας, της σχετικής νομοθετικής πρότασης την επόμενη εβδομάδα θα σταλεί στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για περαιτέρω διαπραγματεύσεις και ελπίζω να ευοδοθούν ώστε η νομική βάση να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2018. Επίσης, έχουμε ένα κοινό πλαίσιο με τη δήλωση της αποστολής, τις και το χάρτη. Τέταρτη διαφάνεια, ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της πρωτοβουλίας. Θα έχουμε δύο ε, συμπληρωματικούς άξονες, τον αθελετισμό και τη μαθητεία. Επίσης έχουμε συμβατικές σχέσεις ε, για τις, ε, για τις μαθητείες, ενώ ο εθελοντισμός είναι πιο ανοιχτό. Είναι ανοιχτός, ε, ανοιχτό το πρόγραμμα σε νέους 18 με 30 ετών και η διάρκεια από 2 με 12 μήνες. Είναι ευρύ το φάσμα των δραστηριοτήτων αλληλεγγύης και το γεωγραφικό επίσης πεδίο εφαρμογή που κατά κανόνα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά μπορεί να επεκταθεί. Επίσης, έχουμε την ροή εργασία. ξεκινάει από την εγγραφή στο σώμα, την ε, υποβολή αιτήσεων, την τοποθέτηση και τη συμμετοχή σε ένα δίκτυο που θα ε, στελεχώνεται και στο, στην πορεία του προγράμματος. Επίσης, εδώ έχουμε τα πλεονεκτήματα για, για τους ε, συμμετέχοντες και για τις οργανώσεις. Θέλουμε να κάνουμε μια αντιστοίχηση των νέων με, τις, με τους διάφορους φορείς, προκειμένου να αυξήσουμε τις συνέργειες μεταξύ των διαφόρων μέσων και μηχανισμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ έχουμε τα διάφορα προγράμματα χρηματοδότησης στην 8η διαφάνεια που ήδη ε, εμπλέκονται και σας είπα ποια είναι η χρηματοδότηση από την ΚΑΠ. Θέλουμε να τη χρησιμοποιήσουμε για να έχουμε κοινή διαχείριση. Για παράδειγμα, στα πλαίσια του πρώτου πυλώνα στο στο πρόγραμμα για το διανομή τροφίμων στα σχολεία μπορούν εκεί να συμμετέχουν οι εθελοντές αλλά και σε δραστηριότητες διαφήμισης ή ενημέρωσης. Αυτό στον πρώτο πυλώνα. Στο δεύτερο πυλώνα έχουμε διάφορα μέτρα σε προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης. Και εκεί θα μπορούσαν να συμμετέχουν οι εθελοντές του Σώματος Αλληλεγγύης για την διαχείριση διαφόρων προγραμμάτων. Το Λίντερ θα διαδραματίσει κέριο ρόλο στην εφαρμογή των πρωτοβουλειών του Σώματος Αλληλεγγύης, ιδιαίτερα στην Ήπεθρο. Και για να ολοκληρώσω, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δώσατε να σας παρουσιάσω εν συντομία την πρωτοβουλία αυτή. Προσπάθησα να σας κάνω μια σύντομη προφορική επισκόπηση των στόχων του Ευρωπαϊκού Σώματος Ελίγης και να επιστήσω την προσοχή σας ε, ε, στη συνάφεια μερικών δραστηριοτήτων του Σώματος Ελίγης και ε, το, της γεωργίας και της γεωργικής ανάπτυξης. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Έχουν ζητήσει το λόγο τόσοι πολλοί συνάδελφοι που με οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν πρόκειται να ικανοποιήσουμε όλη την περιέργεια όλων ή να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ένα λεπτό στον καθένα θα δώσω, γιατί έχουμε και το διαρθρωμένο διάλογο στο πρόγραμμα. Αν χρειαστεί, ίσως, θα ίσως κάποια στιγμή στο μέλλον θα πρέπει να οργανώσουμε νέα συνάντηση για να επανέλθουμε στο θέμα αυτό. Ένα λεπτό λοιπόν ο καθένας, ο κύριος Φέντερλε. Φέντερλε, παρακαλώ. Θα αποσύρω το χρόνο αγόρευσης. Θα μιλήσω για το επόμενο σημείο της ε, οδηγίας. Oui, oui, merci, euh, Président. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, διάβασα προσεκτικά την αναγκή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Σαμαριλεγγύη. Πολλέ πτυχέ ε, με προβλημάτισαν και με ενδιαφέρουν. Θα ήθελα τελικά να μου πείτε κάτι για τη σύγχυση. Θα πρέπει να είναι νόμιμο κάτοικο υπήκο των κρατών τη Ευρωπαϊκή Ένωση ο νέο εθελοντή. Αλλά όχι μόνο. Αναφέρεται ότι μπορεί να ζητήσει ε, και κάποιο που είναι από την Τουρκία ή από, την, ε, από το Φύρομ Πώς ένα πρόγραμμα απασχόλησης ή εθελοντικό μπορεί να προσλαμβάνει ανθρώπους από μη ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η πρωτοβουλία θα μπορούσε να είναι πρώτη χρηματοδοτούμενη από τα εργαλεία που υπάρχουν. Πια το FEDER και το LEADER φαντάζομαι δεν πιστεύω ότι αυτά τα προγράμματα του δεύτερου πυλώνα τη κοινή αγροτική πολιτική είναι πιο καλά για να βοηθήσουν εκείνου που εργάζονται στην Ήπεθρο και του αγρότε. Αναφέρεται ότι μπορούν να βοηθήσουν τα προγράμματα στην υποδοχή και ένταξη των προσφύγων ή καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων. Δεν καταλαβαίνω πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Γιατί η ανάπτυξη τη Ήπεθρου ε, να ασχολείται με αυτό το θέμα. Σα ευχαριστώ εκ των προτέρων που θα με διαφωτίσετε από αυτού. Ε, Σας ευχαριστώ. Έχω τρεις ερωτήσεις. Καταρχήν, θα πρέπει να γίνει διάκριση των ε, δράσεων στις οποίες θα συμμετέχουν αυτοί οι εθελοντές. Ε, επίσης, ε, τι δραστηριότητες θα ασκούν οι μισθωτοί αυτό του σώματος αλληλεγγύης και ποιο θα είναι το επίπεδο των μισθών των απασχολουμένων σε αυτό το σώμα αλληλεγγύης. Γιατί να μην χρησιμοποιηθεί το σώμα ώστε να μειωθεί το μισθολογικό κόστος χρησιμοποιώντας ε, το επισφαλές εργατικό δυναμικό και εκμεταλλευόμενο στους νέους. Θα ήθελα να διευκρινιστούν λοιπόν αυτά τα τρία σημεία. Ευχαριστώ κύριο Φλάναγκαν. Ε, ε. Ευχαριστώ πολύ. Ενδιαφέρουσα η παρουσίασή σας. Πάνω στα όσα υπόθηκαν τι είδους αμοιβή θα δίδεται. Λέτε είναι για αυτούς που είναι ανάμεσα στα 18 και 30. Η μητέρα μου και ο πατέρα μου είχαν 5-6 ε, παιδιά μέχρι να γίνουν 30. Πώς θα επιβιώσουν αυτοί οι άνθρωποι. Θα είναι αυτοί που έχουν αρκετά χρήματα για να μπορούν να είναι θελοντές. Γιατί η μαμά και ο μπαμπάς έχουν χρήματα να τους θρέψουν. Ένας απλός καθημερινός άνθρωπος πώς θα επιβιώσει σαν εθελοντής Πόσο θα αξίζει για τον κόσμο αυτό. Θα μπορούν να φάνε ένα πιάτο φαΐ, να πληρώσουν τον νίκη. Ξέρω εγώ. Περί πρόκειται. Ποιον, καλύπτει. Ευχαριστώ Κύριε Γιλέρα. Κύριε Επίτροπε, εγώ οφείλω να ομολογήσω ότι έμεινα καταθουσιασμένη από την πρωτοβουλία αυτή. Θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και πιστεύω ότι μπορεί να προσφέρει αυτή την αξία της αλληλεγγύης. Και γι' αυτό είναι και πολύ ενδιαφέρουσα η πρωτοβουλία και πολύ ελκυστική για τους νέους κατά τη γνώμη μου. Έχω κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις. Εμείς στην Ισπανία έχουμε ένα αντίστοιχο σύστημα πολιτικής προστασίας. Κάτι παρόμοιο με αυτό που προτείνει και το Σώμα Αλληλεγγύης, από ό,τι κατάλαβα. Έχω όμως μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Όταν μας είπε είπατε σε ποιες δραστηριότητες συμμετέχει η Γεωργία μαζί με άλλους τομείς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε τι ακριβώς δραστηριότητες, γιατί φαντάζομαι αυτό γίνεται στα πλαίσια των ομάδων Leader για την αγροτική ανάπτυξη ή και για κάποιες άλλες πρωτοβουλίες. Σε τι είδους πρωτοβουλίες γεωργίας μπορούν να συμμετέχουν οι νέοι αυτοί. Και τα κράτη-μέλη οφείλουν να ε, θεσπίσουν αυτό το μητρό ή θα γίνεται η διαχείριση του σώματος αλληλεγγύης σε κεντρικό ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα ήθελα αυτό να διευκρινίσω γιατί το θέμα είναι πολύ σημαντικό και η πρωτοβουλία πραγματικά αξιέπαινει. Ο Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να πω παρόμοια με αυτά που είπε η Κλάρα Αγγιλέρα. Η πρωτοβουλία θεωρώ είναι ότι είναι, αρκετά ελκυστική. Επιτρέπει στους νέους, στους νέους Ευρωπαίους δεν είναι υποχρέωση, είναι θελοντική πράξη, έτσι δεν είναι. Τους επιτρέπει να συναντηθούν, ε, να ανήκουν σε μια κοινότητα. Λοιπόν, είναι πιστεύω αυτό σημαντικό, τους ενώνει, επιτρέπει στους Ευρωπαίους να συναντώνται σε κάποια χώρα, να ενώνονται μέσω κάποιας ε, δραστηριότητας, ε, να ανταλλάξουν απόψεις, να γνωριστούν, να δεχτούν τις διαφορές και να συμβάλλουν, πιστεύω, στην οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής Υπήρου που, και να την αντιληφθούν. Λοιπόν, είναι ενδιαφέρον. Δεν μιλάμε για την αμοιβή από ό,τι κατάλαβα από το κείμενο. Περισσότερο την ανάληψη των, του, το κόστος ταξιδίου, ασφάλεια, διαμονή κλπ. Ε, για να μπορέσουν να συναντηθούν. Λοιπόν, στο γεωργικό κομμάτι, εσείς επίπεδο, στο πεδίο της γεωργίας, τι έχετε παρατηρήσει. Ε, υπάρχει ζήτηση. Και αν ναι, για ποιο τομέα έχετε κάποια στοιχεία να μας δώσετε, να κάνουμε κάποια αξιολόγηση πέρα από τη συνάντηση των πολιτισμών και της κουλτούρας υπάρχει και το θέμα των διαφόρων επαγγελμάτων της Γεωργίας. Ήταν ενδιαφέρον να δούμε τι είδους δραστηριότητε ενδιαφέρουν τους νέους. Και αυτό θα μπορούσε να δώσει κάποια στοιχεία για ανάλυση και να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα, πάρουμε μια εικόνα. Κύριος ε, ήθελα να θέσω ερωτήσεις που ήδη ετέθησαν. Νομίζω ότι με κάλυψαν. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ θετικό να γίνονται τέτοιες ε, προσφορές στους νέους. Εδώ και 20 χρόνια υπάρχει η εθελοντική υπηρεσία, η ευρωπαϊκή. Οπότε πώς διαφοροποιείται αυτό το καινούριο για τους νέους, γιατί η γέννηση αυτή του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης ε, προχώρησε πολύ γρήγορα, ε, οι οργανώσεις των νέων δεν ήξεραν τίποτε για την έλευση αυτού του νέου σώματος. Μια νυχτή σχεδόν παρουσιάστηκε και πολλοί ε, απόρρισαν γιατί να μην χρησιμοποιηθεί ε, το Ευρωπαϊκό, ευρωπαϊκό Ευρωπαϊκός Οργανισμός που έχει εμπειρία 20 χρόνων και έγινε κάτι καινούριο. Και εγώ δύο διευκρινιστικές ερωτήσεις. Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση, μεμονωμένες επιχειρήσεις ή κοινοφελείς οργανισμοί, σύλλογοι ή περιοχές leader και πώς κατανέμονται τα κονδύλια. Υπάρχει μια εθνική ποσόστοση ή θα είναι ένα ευρωπαϊκό ταμείο το οποίο με συγκεκριμένη κλίδα κατανέμεται στα κράτη-μέλη. Πώς θα λειτουργήσει στη Γερμανία για παράδειγμα, διότι υπάρχει νοοτροπία ότι όταν υπάρχουν χρήματα όλοι θα πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν. Κυρία Ράς, έχω κι εγώ μια ερώτηση. Διάβασα στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι έχουμε δύο άξονες, ε, τον ε, εθελοντικό και τον επαγγελματικό. Φαντάζομαι ότι και οι εθελοντές θα έχουν κάποια μερίσια αποζημίωση, στέγη, αλλά αυτοί που δεν παρακολουθούν ε, κάποια κατάρτιση, άσκηση, αλλά ε, απασχολούνται, οι συμβάσει θα διέπονται ή θα συνάπτουν σε εθνικό επίπεδο ή σε ευρωπαϊκό. Και ποιο θα χρηματοδοτήσει την πρωτοβουλία αυτή, Γιατί είναι, θα είναι το leader, κανένα άλλο πρόγραμμα. Πώ θα χρηματοδοτηθούν αυτέ οι συμβάσει και το σώμα γενικώ. Ο πρόεδρο. Η ιδέα είναι πολύ ωραία, κυρίε και κύριοι. Ο κύριο Χόγκαν μας παρουσίασε αυτή την ε, ιδέα του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Βέβαια, η πραγματικότητα δεν είναι θεωρία. Θα πρέπει να δούμε πώς εμπράκτος εφαρμόζεται το πρόγραμμα. Και, για παράδειγμα, ένας φοιτητής μπορεί να απασχοληθεί στη γεωργική εκμετάλλευση του κυρίου Γιάρ και να αξιοποιήσει την εμπειρία που θα χρησιμοποιήσει εκεί ή σε μια άλλη γεωργική εκμετάλλευση αν θεωρήσουμε ότι είναι κατάρτιση, άσκηση. Ωραία, σε μια γεωργική εκμετάλλευση έχει πολλά να μάθει ένα φοιτητή, α πούμε. Είπα, η γεωργική εκμετάλλευση του γύρου Γιάρ θα μπορούσε να είναι το Α ή του Β. Έτσι, τυχαία χρησιμοποιήσει αυτό το παράδειγμα. Πώ θα διαθετηθούν όλα αυτά. Ο Επίτροπο έχει το λόγο για να απαντήσει. you, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλου εκείνου που έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για το ζήτημα. Το είδα τι ερωτήσει που έκαναν. Πρώτα απ' όλα, ε, είναι σημαντικό οι λεπτομέρειες που περιέχονται στην πρωτοβουλία θα πρέπει να αποκαλυφθούν. Και αυτό μέσω των συζητήσεων που θα γίνουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την επόμενη εβδομάδα. Και οι συνομοθέτες θα πρέπει να θεσπίσουν το κατάλληλο νομικό πλαίσιο. Ίσως, Πρόεδρε, την επόμενη εβδομάδα στην Αγκρή να δώσω εγώ τις λεπτομέρειες που διαθέτω μετά τη συνάντηση που θα έχουμε στην Κομισιόν την επόμενη εβδομάδα. Περισσότερες πληροφορίες από ό,τι μπορούσα να δώσω τώρα. Κοιτάξτε, είναι ένα πρόγραμμα αυτό που στρέφεται προς τους εθελοντές. Ανακοινώθηκε σαν πρωτοβουλία από τον πρόεδρο, τον Ζαν Κλοντ Γιούγκερ, στη δήλωσή του τον περασμένο Σεπτέμβριο την κατάσταση της Ενώσεως. Η πρόθεσή του ήταν να υποβάλει προτάσεις που θα επιτρέπουν στους νέους να μπορούν να συμμετέχουν με τον πληρέστερο δυνατό τρόπο σε διάφορα εγχειρήματα που είναι φιλικά προς την κοινωνία, εθελοντικά βασικά. Δεν θέλουμε να προσλαμβάνουμε φθηνό εργατικό δυναμικό για να συμπιέσουν προ τα κάτω τι αμοιβέ. Δεν είναι που δεν είναι αυτό ο σκοπό πρωτοβουλία. Θέλουμε να δημιουργήσουμε προστιθέμενη αξία μέσω αλληλεγγύη σε κάποιε περιστάσει που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Που αφορά τη μετανάστευση, του πρόσφυγε, τι φυσικέ καταστροφέ, είτε είναι πυρκαγιέ, είτε είναι σεισμοί, οτιδήποτε. Αυτό θεωρήθηκε ότι είναι μια ευκαιρία να μαζευτούν οι άνθρωποι στα πλαίσια τη αλληλεγγύη και να κάνουν κάτι. Και αυτό είναι πολύ καλό. Το πιλωτικό πρόγραμμα μέχρι τώρα επέτρεψε ευελιξία για τα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες. Αν επιθυμούν εντελώς εθελοντικά να συμμετέχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, αν θέλουν να διαθέσουν ένα μικρό ποσό, όπως είδατε στο πιλωτικό πρόγραμμα, εγώ έδωσα 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό δεν φαίνεται και πολύ μεγάλο ποσό και δεν νομίζω ότι θα θεωρήσουν ότι είναι επιζήμιο ή ότι είναι πολύ ακριβό εκείνοι που είναι εναντίον του προγράμματο. Εάν όμω είναι ελκυστικό, αν έχει αποτελέσματα το πρόγραμμα, μπορούμε να έχουμε περισσότερα χρήματα στο μέλλον. Αυτό θα το αποφασίσετε και εσεί στο μέλλον. Ο δεύτερος, η χρηματοδότηση του δεύτερου πυλώνα υπάρχει πάντα για την ευελιξία όσον αφορά την ανάπτυξη τη υπαίθρου και για τι φυσικέ καταστροφέ. Ούτω ή άλλω. Και έχουμε άλλη μια διάσταση που προσθέτουμε. Για εκείνου που θέλουν να δηλώσουν εθελοντέ για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων των προβλημάτων που να είναι φυσικέ καταστροφέ. Οι εφαρμοστικοί φορεί θα είναι οι εθνικοί φορεί του Erasmus Συν, ε, Erasmus Plus. Δεν δημιουργούμε νέε δομέ. Και διάφορε φορεί για τα οπτικοκουστικά, ε, παιδεία κλπ. Η αρμόδια γενική διεύθυνση. Όλε οι γενικέ διευθύνσει και η Γενική Διεύθυνση Γεωργία θα ε, κινηθούν μέσω των υφισταμένων δομών. Δεν δημιουργούμε κάποια ξεχωριστή δομή για το συγκεκριμένο θέμα. Άρα είναι στα πλαίσια της κοινή διαχείρισης. Το Erasmus Plus θα δώσει 58 εκατομμύρια ευρώ. Το πρόγραμμα απασχόλησης κοινωνικής καινοτομίας θα δώσει 5,2 εκατομμύρια. Το LIFE 2 εκατομμύρια. Η Ευρώπη για τους πολίτες 3,5 εκατομμύρια. Άσυλο, μετανάστευση και ένταξη 9,6 εκατομμύρια. Κοινή αγροτική πολιτική 1,8 εκατομμύρια. Έτσι έχετε μια εικόνα του ευρέω φάσματο ε, τομέων που συμμετέχουν και ποιο είναι ο σκοπό. Όπω είπα, Πρόεδρε, καταλαβαίνω μεν ότι θέλει ο κόσμο πληροφορίε και καλά κάνει. Η παρέμβασή μου εδώ έχει σαν στόχο να σα δώσω μια έτσι εικόνα, να σα πω τι γνωρίζω μέχρι τώρα αφορά το πιλωτικό πρόγραμμα θα κάνω ό,τι μπορώ να σα δώσω περισσότερε πληροφορίε την επόμενη εβδομάδα που θα τι διαθέτω. Και αν θέλετε να θέσετε και άλλε ερωτήσει σε μελλοντική συνάντηση, μπορώ να απαντήσω. Θα απαντηθούν το μεταξύ και πολλέ ερωτήσει σα από τι πληροφορίε θα πάρετε την επόμενη εβδομάδα. Θα μπορέσετε επίση ε, να δείτε και τι νομικέ συνέπειε θα υπάρξουν ε, κατά τη διάρκεια τη νομοθετική διαδικασία, που ελπίζουμε αυτή να ολοκληρωθεί από τώρα μέχρι το τέλο του έτου. Πρόεδρε, πρόεδρε έχουμε ελάχιστη εμπειρία. Διότι τους πρώτους ανθρώπους τους ε, προσλάβαμε, αν θέλετε, αρχές Μαρτίου ήρθαν. Πάντως, ε, χαίρομαι που μας ε, είπατε ότι θα μας ενημερώνετε γενικώ για την πορεία των συζητήσεων και σε άλλες, σε άλλες επιτροπές του Κοινοβουλίου. Ωραία, ολοκληρώσαμε το πρώτο θέμα που ήταν προκαταρκτική συζήτηση μετά την παρουσίαση για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Δεύτερο θέμα είναι ο διαρθρωμένος διάλογος στα πλαίσια ε, της διοργανικής συμφωνίας που διέπει τις ε, σχέσεις και Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου και γίνεται πάντα στο πρώτο εξάμεινο κάθε Ε, γίνεται τόσο ο διάλογο διάλογος μεταξύ των ε, επιμέρους κοινοβουλευτικών επιτροπών και των επιτρόπων που έχουν χαρτοφυλάκιο που εμπιτήσει ενδιαφέροντα των επιτροπών. Ε, στα πλαίσια του διαλόγου θα δούμε πώς δρομολογούνται οι δραστηριότητες του προγράμματος εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2015 και θα ε, γίνει και μια παρουσίαση των ε, προτεραιοτήτων για το 2018, για το επόμενο έτος δηλαδή, για να μπορέσουμε και εμείς να συμβάλλουμε τις προτάσεις μας στη διαμόρφωση του μελλοντικού προγράμματος εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σκεφτήκαμε ότι για το διερθωμένο διάλογο ο καλύτερο τρόπο είναι να υποβάλουμε εκ των προτέρων ερωτήσει για να προετοιμαστεί ο Επιτροπό και σα ευχαριστώ θερμά γιατί υποβάλλατε πραγματικά πλειάδα ερωτήσεων. Καλύπτουν αυτές ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Έτσι μπόρεσε και ο Επίτροπος να ενημερωθεί για την γενική κατεύθυνση του προβληματισμού μας. και να προετοιμαστεί. Οπότε αυτές τις ερωτήσεις θα μπορούσαμε εν συντομία να τις υποβάλουμε και σήμερα στην συζήτηση που θα έχουμε με τον Επίτροπο. Θα δώσω πρώτα το λόγο στον Επίτροπο Χόγκαν, μετά στους συντονιστές μας. Ε, θα ακούσουμε κατόπιν τις απαντήσεις ε, του Επιτρόπου στους συντονιστές και θα περάσουμε στο δεύτερο γύρο με τις ερωτήσεις των υπόλοιπων Ευρωβουλευτών πολύ σημαντικό το θέμα του διαρθρωμένου διαλόγου, χρονοβόρο. Γι' αυτό και σας δίνω μέσω το λόγο κύριε Επίτροπε. Αυτές ε, οι περιστάσεις είναι χρήσιμες για να συζητήσουμε αμοιβαία σημαντικά θέματα. Μπορεί να έχουμε διαφορετικές απόψεις καμιά φορά σχετικά με το τι πρέπει να γίνει, αλλά πρέπει να συζητάμε. Αυτή τη φορά μου δώσατε πάνω από 40 γραπτές ερωτήσεις και απάντησα. Ελπίζω ότι ελάβατε ήδη τις απαντήσεις και είναι χρήσιμες. Και απόψε είμαστε στο μέσο της εντολής της ε, Κομισιόν. Το πρώτο μέρος της εντολής αφοσιώθηκε στην αντιμετώπιση του ρωσικού εμπάργου, τις πτωτικές τιμές, ιδιαίτερα στα γαλακτοκομικά και το χείριο, την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ και αν υπήρχε επάρκεια των διαθέσιμων μηχανισμών για να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες της αγοράς. Και υπήρξε πρόσθετη δημοσιονομική στήριξη λόγω της ε, οξύτητας της κρίσης εκεί όπου υπήρχε ανάγκη. Και με τις προτάσεις στο πολυνομοσχέδιο και την ε, κατεξουσιοδότηση πράξη για την οικολογική διάσταση της αγοράς, ε, χαίρομαι που επετεύχθη πρόοδος και στο μέλλον θα επιτευχθεί και άλλη πρόοδος. Εκτιμώ ιδιαίτερα την ταχύτητα αντιμετώπισης από πλευρά σας του πολυνομοσχεδίου, του και συγχαίρω τους ε, ε, εισηγητές. Ε, εργαστήκατε στα πλαίσια των προθεσμιών και καλό είναι να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα πριν από το διακοπές του καλοκαιριού επιστονικής προεδρίας. Εσείς το περιοδικό του Κοινοβουλίου ε, αναδείξατε κάποιες προτεραιότητες και συμφωνώ με την προτεραιότητα που δόθηκε στο έργο αυτής της Επιτροπής. Πιστεύω ότι εντοπίσατε τις μεγάλες προκλήσεις των επόμενων δυόμιση ετών ε, στα πλαίσια της ΚΑΠ μετά το 2020, τον προϋπολογισμό για την ΚΑΠ και το πλαίσιο ε, του πολιετούς ε, πλαισίου. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ασφάλεια τροφίμων και ποιότητα τροφίμων. Αυτά, ε, ορισμένα θέματα επηρεάστηκαν από την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει. Τώρα θα πρέπει να δούμε πώς, τι τροπή θα πάρουν αυτές οι διαπραγματεύσεις. Το πιο θετικό αποτέλεσμα εις ό,τι αφορά την ε, γεωργία και τα τρόφιμα είναι να υπάρχει μια εμπορική σχέση που θα προστατεύει τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Βλέπε πρόσβαση στην αγορά ε, θα έχουμε πολλές ευκαιρίες να τα συζητήσουμε όλα αυτά όταν αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις τον Ιούνιο. Τέτοια εποχή πέρσι είχαμε θετικές εξελίξεις κύριε Πρόεδρε σε ό,τι αφορά τη βελτίωση κάποιων τιμών αγοράς αλλά δεν θεωρούμε τίποτε δεδομένο. Η κατάσταση εξακολουθεί να είναι εύθραυστη. Η Κομισιόν αξιοποίησε πλήρως τα, τους μηχανισμούς που διαθέτει στα πλαίσια της κοινή οργάνωσης της αγοράς και χαίρομαι για την υποστήριξη που δώσατε στις προσπάθειες της ε, Κομισιόν. Ο πρόεδρος της Κομισιόν επίσης δεσμεύτηκε ε, υπέρ του μέλλοντος της ΚΑΠ αργότερα φέτος. Ε, μετά από τη δέσμευση κάναμε ανακοίνωση, μετά από δημόσιες διαβουλεύσεις και είχαμε εκατοντάδες χιλιάδες απαντήσεις. Ε, βέβαια εξακολουθούν να απαντούν στα πλαίσια και να, αυτής, αυτών των διαβουλεύσεων. Ενθαρρύνουμε υψηλό επίπεδο συμμετοχής και από αγρότες και μη αγρότες. Η πρώτη ανάλυση των απαντήσεων δείχνουν ότι ε, πολλοί ε, συμφωνούν. Ε, αυτές οι καμπάνιες δεν είναι κάτι το καινούριο. Εμείς ε, πήραμε πάρα πολλές απόψεις, ένα ευρύ φάσμα από πάρα πολύ ευρύ φάσμα εμπλεκομένων. Ε, θα αναλυθούν αυτές οι απαντήσεις και θα γίνει στις Βρυξέλλες στις 7 Ιουλίου μια ε, διάσκεψη εμπλεκομένων. Ελπίζω να συμμετάσχετε και κι εσείς όπως και άλλοι εμπλεκόμενοι στις Βρυξέλλες. Αυτό θα είναι ορόσημο μεταξύ άλλων ε, προς την ανακοίνωση της Κομισιόν. Πρόθεση της Κομισιόν είναι η ανακοίνωση να ε, υιοθετηθεί μέχρι το τέλος του έτους θα πρέπει να βεβαιωθούμε για την βιωσιμότητα της παραγωγής, την ανθεκτικότητα των παραγωγών ε, είναι πολύ σημαντικό η καινοτομία και η τεχνολογία να μπει στην γεωργία και στα, στην τεχνολογία των τροφίμων. Πολλές φορές χρειάζονται απλουστεύσεις. Οι νέες τεχνολογίες θα μειώσουν τις επιθεωρήσεις επιτόπου. Ε, πολλές φορές χρησιμοποιούνται δωρεάν δεδομένα από δορυφόρους στα πλαίσια του προγράμματος Κοπέρνικος και στο στο εγγύς μέλλον πολλοί επιτόπιοι έλεγχοι θα αντικατασταθούν από δορυφορικούς. Αυτό είναι στα σχέδιά μου. Το Ευρωπαϊκός Οργανισμός για το Διάστημα επίσης θα μας δώσει πολλά χρήσιμα στοιχεία και μέσα για να δούμε ε, δορυφορικά δεδομένα για τους δικούς μας ε, σκοπούς. Επίσης υπάρχει πιλωτικό σχέδιο για ψηφιακά εργαλεία, ένα κονσόρσιουμ που αποτελείται από εθνικές διοικήσεις θα υποστηριχθεί για να υπάρξει ένα σύστημα ΩΣΔΕ στο μέλλον που δεν θα επιτρέπει μόνο τη διαχείριση των πληρωμών αλλά θα προβλέπει και για κλιματικά ε, δεδομένα στη Γεωργία. Δεν θα πρέπει να περιμένουμε την, πρώτη, την επόμενη αναθεώρηση της ΚΑΠ για να κάνουμε αυτές τις καινοτομίες. Πρέπει να δουλέψουμε γρήγορα. Ε, υπάρχει και ένα άλλο θέμα που είναι οι αθέμητες εμπορικές πρακτικές και συμφωνώ με τις απόψεις που εκφράσατε και με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σε σχέση με την τροφική αλυσίδα. Θα πρέπει να υπάρχει δικαιοσύνη για τους παραγωγούς, ούτως ώστε να έχουμε βιωσιμότητα, επιβίωση των γεωργών. Ε, αλλιώς δεν θα υπάρχει γεωργικός τομέας. Τώρα εργαζόμεθα για να δούμε τα θέματα της ε, διαφάνειας της αγοράς, τις αθέμινες πρακτικές, τη συνεργασία των ε, παραγωγών ε, και γνωρίζω ότι εσείς ε, ε, ασχοληθήκατε πάρα πολύ στα πλαίσια του πολυνομοσχεδίου για όλα αυτά. Η Κομισιόν τώρα κάνει προπαρασκευαστικό έργο για να διασφαλίσει ότι η περαιτέρω πρωτοβουλία μας θα αντιμετωπίσει και την προϋπόθεση που τίθεται για την καλύτερη νομοθεσία. Θα συζητήσουμε για τους όρους της, και τις προϋποθέσεις της αγοράς, ε, γενικά θα ήθελα να αναφερθώ και στη κατάργηση των ποσοστώσεων ζάχαρης. Το είχαμε πει εδώ και πολύ καιρό και τώρα έχουμε κάνει προετοιμασία για να τελειώσει αυτό το καθεστώς. Ε, προβλέπεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θα γίνει μακροπρόθεσμα εξαγωγέα ζάχαρης λαμβάνοντας υπόψη πρόσθετες ευκαιρίες της αγοράς γιατί αυξάνεται παγκόσμια η θα επηρεαστεί βέβαια και η ε, αστάθεια των τιμών ε, θετικά. η Θα παρακολουθηθεί η αγορά και στο μέλλον, θα υπάρξει παρατηρητήριο για τη ζάχαρη ούτως ώστε να υπάρχει μέγιστη διαφάνεια και ενημέρωση της αγοράς ούτως ώστε να λαμβάνονται σωστές αποφάσεις. Σταματώ στο σημείο αυτό για να ακούσουμε τις ερωτήσεις και ελπίζω ότι θα συμπληρώσω τις γραπτές μου απαντήσεις ε, με βάση τις ερωτήσεις που ήδη μου στείλατε. Όπως ε, είπα, θα δώσω πρώτα το λόγο στους συντονιστές για δύο λεπτά θα ακούσουμε κατόπιν τις απαντήσεις ε, του Επιτρόπου και θα ακολουθήσει δεύτερος γύρος ερώτα-απαντήσεων ανάλογα με το πόσο χρόνο θα έχουμε στη διάθεσή μας. Ο κύριος Νταντά που καθιστά σήμερα τον κύριο Αλμπερντές. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, ο Αλμπερντές, ο συντονιστής μας, δεν μπόρεσε να παραστεί και μου ζήτησε να να σας πω ότι ζητά συγγνώμη για την απουσία του. Θέλω να φέρω σε τρία σημεία. Σε σχέση με αυτά που είπατε και τις πρόσφατες ε, δηλώσεις που έγιναν. Ξεκινήσατε, όπως είπατε, μια συζήτηση. Αυτή αφορά το μέλλον της κοινή αγροτικής πολιτικής. Πολλοί έχουν ασχοληθεί με τη συζήτηση αυτή, κυρίως έχουν συμβάλει οι γεωργοί και πολλοί άλλοι όμως έχουν τοποθετηθεί. Καμιά φορά αντιπροσωπεύονται συγκεκριμένα συμφέροντα, καμιά φορά οι πολίτε. Και καμιά φορά μεταξύ των συμφερόντων των συγκεκριμένων και οι πολίτε. Γίναν κάποιε αναφορέ. Σύμφωνα με τι οποίε αυτά τα χρήματα που πηγαίνουν στου γεωργού τελικά αμείβουν ε, ειδικέ αποστολέ περιβάλλοντο, περιβαλλοντικέ. Έχει αλλάξει η νοοτροπία των γεωργών και οι τεχνικέ που χρησιμοποιούν και αντιλαμβάνονται ότι η προστασία των γεών από την αλλαγή του κλίματος είναι σημαντικός παράγων. Όμως θα πρέπει να επενθυμίσουμε κάτι άλλο. Και ξέρω, θέλω να ξέρω ποια είναι η απόψή σας. Ότι η κοινή αγροτική πολιτική κυρίως προσπαθεί να πετύχει μια οικονομική ισορροπία στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Η κατάσταση που αντιμετωπίσαμε το 2015 και το 2016 μας κατέδειξε τον έφραστο χαρακτήρα του τομέα των εκμεταλλεύσεων. Η ισχύ στο γαλακτοκομικό τομέα δεν έχει βγει ακόμα από την κρίση και έχετε ακόμα στα χέρια σας τόνους ε, γάλακτος σε σκόνη που είναι κάτι αρνητικό για την ευρωπαϊκή αγορά. Το 2016 είδαμε ότι οι κλιματολογικές συνθήκες διετάραξαν το εισόδημα ε, των καλλιεργητών δημητριακών και σε πολλές ευρωπαϊκές περιοχές, σε χώρες ευρωπαϊκές βλέπουμε ότι υπήρξαν κάποια φαινόμενα ακραία καιρικά που είδαν, έγιναν τον Απρίλιο και τον Μάιο και αυτά τα καιρικά φαινόμενα ε, θα επηρεάσουν τα εισοδήματα των γεωργών. Λοιπόν, λοιπόν, αν δεν υπάρξει μεταρρύθμιση δεν θα υπάρχει πλέον γεωργία. Θα πρέπει να επενθυμίσουμε στην κοινή γνώμη ότι η κοινή αγροτική πολιτική έχει ουσιαστικά μια βάση οικονομικής, προστατεύει την οικονομία του τομέα. Μπόρεσα να δω ε, πόσο προβληματισμένη είναι η Γεωργοί στη χώρα μου στις τελευταίες εβδομάδες. Η απελπισία τους ε, ξεπερνά αυτό που φανταζόμουν και η ανησυχία τους. Πολύ συχνά η γάλακτοπαραγωγή, θέτουν αυτή την ερώτηση. Τι γίνεται με τα αποθέματα γάλακτος ε, σε σκόνη που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς αυτά θα διατεθούν, γιατί απειλούν τη σταθερότητα των τιμών. Το θέμα είναι πώς θα το διαθέσουμε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να μην επηρεάσουμε τις ε, τιμές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αν διατεθούν αυτά τα θέματα γάλακτος σε σκόνη στην ευρωπαϊκή αγορά θα ρίξουν πολύ τις τιμές. Ευχαριστώ κύριος ε, Αντριέ. Ευχαριστώ. Εγώ ζήτησα το λόγο για την πρόταση Omnibus και τι συνέχεια θα δοθεί. Ξεκίνησε κάπως και ο κύριος Δαντά με αυτό το θέμα στην τελευταία μας ψηφοφορία στην Επιτροπή Γεωργίας. Ξεπεράσαμε κάπως ε, το πλαίσιο που μας είχατε θέσει. Ε, ήταν πάντως ξεκάθαρο το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Εγώ λοιπόν θα ήθελα να σταθώ στις ε, ουσιαστικές ε, τροπολογίες που προτείναμε στην ενιαία κοινή οργάνωση αγοράς και στις προτάσεις μας για την καταπολέμηση των αθέμητων εμπορικών πρακτικών, τις οποίες ακροθυγώς αναφέρατε κι εσείς. Επίσης ένα άλλο θέμα, ε, διόλου σήμαντο, που αφορά την καλύτερη οργάνωση των παραγωγών και την προσαρμογή όλων των κλάδων στους κανόνες του ανταγωνισμού, ώστε να επιτρέπει καλύτερη οργάνωση. Και επίσης η γενίκευση αυτής της ε, ε, εθελοντικής και έκτακτης διαχείρισης των όγκων των ποσοτήτων σε περίπτωση σοβαρής κρίσης. Στους τριμερείς διαλόγους που θα ακολουθήσουν φαντάζομαι είχατε κάπως ε, προσταθεί αυτή τη θέση της Επιτροπής Γεωργίας. Πώς λοιπόν θα τη λάβετε υπόψη τη συνέχεια των διαπραγματεύσεων και σε ό,τι αφορά τη μελλοντική μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, σε ό,τι αφορά τη, τα θέματα που ζητή, θέσατε εσείς και αυτά που μας προβληματίζουν και τα οικονομικά, δεν θα πρέπει να ενδώσουμε και να δεχτούμε περικοπές ενώπιστων μεταρρυθμίσεων, γιατί έτσι θα σκάψουμε μόνοι μας το λάκκο μας. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε ευρηματικούς και αφάνταστους τρόπους, όχι μόνο να, για να νομιμοποιήσουμε την ΚΑΠ, αλλά να της δώσουμε και νόημα ταυτόχρονα. Επίσης θα πρέπει να βρούμε το σωστό σύνδεσμο μεταξύ της παραγωγής και της κατανάλωσης, με σεβασμό φυσικά της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, όπως είπε και ο κύριος Νταντάν πριν από λίγο. Σε ό,τι αφορά την τροφική αλυσίδα, οι γεωργοί λένε ότι η οικονομία ε, της τροφικής αλυσίδας δεν αρχίζει στο αγρόκτημα και σταματάει στον καταναλωτή, αλλά ξεκινάει από τις τιμές των προϊόντων που χρειάζεται να αγοράσουν για την παραγωγή τους οι καταναλωτές, τα λιπάσματα, τα φυτοφάρμακα, τις ζωοτροφές, τις, τους σπόρους. Γιατί οι γεωργοί λένε, μας ε, μιλάτε μόνο για την αλυσίδα από τον αγρό στο τραπέζι. Αλλά τι γίνεται με τα προϊόντα που οφείλει να αγοράσει ο Γεωργός και αυτά επίσης επηρεάζουν το γεωργικό του εισόδημα και το μειώνουν. Θα πρέπει να επεκτείνουμε λοιπόν την τροφική αλυσίδα και να καλύψουμε και κάποια πρώτερα στάδια από τον αγρό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νίκολσον θέλει το λόγο τώρα ή αργότερα. Εντάξει, τώρα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη που δεν ήμουν εδώ. Ήμουνα στην Ολομέλεια και μιλούσα για τη σπατάλη των τροφίμων. Και θα πρέπει εμείς που συμμετέχουμε στο Κοινοβούλιο και είμαστε δραστηροί θα πρέπει να ειδοποιούμε όταν προσπαθούμε να πρέπει υποτίθεται να είμαστε πανταχού παρόντες. Λοιπόν, έχουμε και άλλες υποχρεώσεις την ίδια χρονική στιγμή. Χαίρομαι που σας αναβλέπω, Επίτροπε. Σας έβλεπα στην τηλεόραση το Σαββατοκύριακο που με πηγαίνατε στο Κάντι Μάλαχαν και βλέπατε τις αγελάδες. Και ήρθε και ο κύριος Μπαρνία και είσαστε σε μια σημαντικότητα υποστολή. Τα λέω μα. Ξέρω ότι είστε ικανότατος πολιτικός και δεν σας ενοχλώ. Μπορείτε να αντέξετε την πίεση και να σταθείτε στα πόδια σας. Γι' αυτό τα λέω αυτά. Μπορείτε, μπορείτε να αποσπάσετε κάτι από τον κύριο Μπαρνιέ παραπάνω για την όλη κατάσταση. Πήγα στο Μπάλμαρο την περασμένη εβδομάδα στο σοου. Είναι μια έκθεση γεωργία στη Βόρεια Ιρλανδία, μεγαλύτερη έκθεση. Και όπου και να πήγαινα και με όσου μιλούσα, με ρωτούσαν τι θα συμβεί. Ποιο θα είναι το μέλλον. Ξέρω ποια είναι η κατάσταση. Τίποτα θα συμβεί όσον αφορά το Brexit πριν τον Οκτώβριο για να τελειώσουν οι γερμανικές εκλογές. Αυτή είναι σκληρή αλήθεια. Αλλά οι απλοί άνθρωποι ε, ακούν αυτά που τους λένε τα ΜΜΕ και κάποιοι πολιτικοί. Τους θα παρουσιάζουν κάποιοι όλα σκοτεινά, θεοσκότεινα, ότι θα συμβούν τα πάντα, θα καταρρεύσουν τα πάντα και δεν θα μείνει τίποτα για κανέναν. Επίτροπε, αυτή είναι η αλήθεια. Δεν ήρθε η ώρα κάποιοι να δουν ποια είναι η πραγματικότητα, να βγει μια ρεαλιστική εικόνα. Θα συμβούν κάποια πράγματα. Ξεκίνησε η μπάλα να ρολάρει. Θα πρέπει να συνεργαστούμε μεταξύ μας. Προς όφελος όλων. Όλων των χωρών μας και των περιοχών μας. Να ωφεληθούν όλοι μακροπρόθεσμα. Όχι μόνο εντός Ευρωπαϊκής Ενώσεως, αλλά και στο Ηνωμένο Βασίλειο όταν αποχωρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο. Ας απαλλαγούμε από όλη τη ρητορική. Μιλούσαν ε, για την τη διπλωματία των μεγαφώνων από την ε, άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Τώρα μιλάνε από την, άλλη... Ε, την πολιτική των μεγαφώνων την άλλη πλευρά της μάχης. Να κάνουμε κάτι επικοδομητικό, να σταματήσουν αυτά. Ξέρω ότι στο επίκεντρο αυτό αλλά είναι ένα από τα μεγάλα μεγάλα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουμε τους επόμενους 12 μήνες. Κυρία Μίλλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κι εγώ έπρεπε να μιλήσω στην Ολομέλεια και καθυστέρησα. Η κοινή πολιτική έχει και την πράσινη διάσταση, το, την οικολογική συνιστόσα, και τη σχετική στρατηγική στην Ευρώπη. Προφανώς μας ενδιαφέρει να μην ε, χάσουμε την εμπιστοσύνη των γεωργών. Οι γεωργοί πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη στην πολιτική. Πρόκειται για την αξιοπιστία μας. Και αν ε, θέλουμε να ε, εφαρμόσουμε, αν εφαρμόσουμε δύο χρόνια το greening, την πράσινη διάσταση και ε, δεν επιτρέπουμε τα, τη συνέχιση των καλλιεργιών των αμιλούχων φυτών, τότε θα έχουμε πρόβλημα. Επίσης, οι online διαβουλεύσεις στο δίκτυο υπάρχουν κάποια αποτελέσματα. Την ε, συμμετοχή των ε, κλάδου που ε, υπέρ της προστασίας της φύσης, πώς την αξιολογείται. Έχουμε πάρα, πολλά, πάρα πολλές ε, παρεμβάσεις από όλες τις μεγάλες χώρες. Πέντε χώρες συμμετείχαν, ε, Ισπανία, Γαλλία, ε, Γερμανία, πέντε από 28. Και έχουμε 285.000 υποστηρικτές της πρωτοβουλίας που ανελήφθη μαζί με την WWF για την προστασία της φύσης. Εσείς αυτή την αξιολόγηση πώς θα ε, διασφαλίσετε ότι αυτά τα μαζικά mail δεν θα ε, υπονομεύσουν την ΚΑΠ στο μέλλον γιατί η online διαβούλευση θα έπρεπε να οδηγήσει σε μια αντικειμενική συζήτηση με πρακτικά αποτελέσματα και λύσεις για τους γεωργούς. Και το τρίτο σημείο που αν με επιτρέπετε ε, στην δική μας την περιφέρεια στη Γερμανία ε, είχαμε πάρα πολλές ε, ζημίες ε, από τον παγετό στα μπέλια και στα εσπεριδοειδή, όπως επίσης και στα κεράσια από 20 μέχρι 70% σε ορισμένες ποικιλίε. Και τώρα συζητούμε στη Γερμανία πώς θα αντιμετωπίσουμε το Ταμείο για την Κρίση και αν μπορούμε ή αν θα πρέπει να το παρουσιάσουμε ως φυσική καταστροφή όπως έκανε η Βάδη Βιρτεμβέργη και έτσι θα πρέπει ε, να παρουσιάσουμε ε, μεγάλη καταστροφή, μεγάλης ε, κλίμακας. Πώς θα προστατεύσουμε τους αγρότες μας και τι πρέπει να κάνουμε εμείς τα κράτη-μέλη ούτως ώστε να δοθούν κάποιες αποζημιώσεις. Αυτές ήταν οι ερωτήσεις μου και σας ευχαριστώ πολύ η κυρία Σένερα που μίλησε και προηγουμένως. Ευχαριστώ. Έχω και εγώ πολλές ερωτήσεις. Κύριε Επίτροπε, είπατε στη Μαδρίτη ότι δεν θα, δεν, δεν θα γίνει πραγματική μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, αλλά απλώς απλούστευση και εξυγχρονισμό τη κοινή γεωρική πολιτική. Και αυτό το άκουσα και από άλλου εκπροσώπου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι ακριβώ εννοείται με εξυγχρονισμό τη κοινή γεωργική πολιτική. Επίση, είπατε ότι συνεχίζονται οι διαβουλεύσει. Πώ γίνονται αυτέ οι διαβουλεύσει, τι απόψει συγκεντρώνεται και από ποιου και τι βαρύτητα δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις ε, απόψεις των ε, αγροτικών επαγγελματικών οργανώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μία άλλη ερώτηση που θα ήθελα να κάνω είναι πώς θα προσεγγίσετε ε, τα προβλήματα που δημιούργησε η απορρίθμιση. Ε, γιατί εξακολουθεί να σοβεί η κρίση στον γαλακτοκομικό τομέα, οι τιμές είναι κάτω του κόστους, ε, ε, χρηματοδοτήθηκε με δημόσια κονδύλια η εθελοντική απόσυρση στο γαλακτοκομικό τομέα, αλλά συνεχίζεται η συζήτηση στην Ισπανία, για παράδειγμα. Ε, ακούστηκε η περίπτωση της γεωργικής εκμετάλλευσης ε, γιατί με 20.000 αγελάδες. Πώς θα προστατεύσετε τους ε, παραγωγούς του γάλακτος από τέτοια προβλήματα. Επίσης, για το θέμα των τιμών, είπατε ότι θα καταργηθούν τόσο λίγο και οι ποσοστό στη ζάχαρη, οπότε αναμένεται μεγάλη διακύμαση των τιμών και μεγάλη αστάθεια και στις τιμές της ζάχαρης. Εξετάζεται σοβαρά το θέμα της ρύθμισης ε, της παραγωγής και της ρύθμισης των αγορών. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χόισλινγκ. Äh, Κύριε Επίτροπε, και εγώ έχω να κάνω κάποιες ερωτήσεις. Ε, είπατε ότι συμμετείχαν ε, πάρα πολλοί ε, και από το περιβάλλον είναι πολλοί δηλαδή αυτοί που ενδιαφέρονται για το περιβάλλον και δεν είναι ενεργοί γεωργοί. Νομίζω ότι αυτοί που εργάζονται στη γεωργία πρέπει να συμμετέχουν στην ε, αναμόρφωση και τη μεταρρύθμιση της ε, ΚΑΠ. Ε, βεβαίως και δεν θέλουμε να ε, περιθωριοποιήσουμε κανέναν. Όλοι θα πρέπει να συμμετέχουν. Για το γάλα, σήμερα ένας μεγάλος ε, συνεταιρισμός στη Γερμανία είπε ότι στα 32 cents ε, μπαίνει όριο, δεν μπορεί να δοθεί παραπάνω. Ε, τώρα μειώνονται οι τιμές για το γάλα. δηλαδή, τι θα γίνει στο μέλλον, και σε ό,τι αφορά τον κανονισμό ε, Omnibus ε, πως θα έπρεπε να προβλέψουμε κάποια μέτρα για την αγορά για να προλάβουμε ε, δυσάρεστες εξελίξεις στο μέλλον. επίσης για τους σπόρους είπατε ότι τα 15 χρόνια διάρκεια δεν παρουσιάζουν πρόβλημα αλλά θα πρέπει να δούμε και τον καρκινογόνο χαρακτήρα ορισμένων ουσιών γιατί υπάρχει μεγάλη επίπτωση στην βιο ε, ε, τελευταία ερώτηση, η δορυφορική παρακολούθηση. Είπατε ότι τώρα υπάρχουν καλύτερες δυνατότητες ε, δορυφορικής παρακολούθησης. Δηλαδή τι θα βελτιωθεί, τι είναι το καλύτερο θα μετράνε το χιλιοστό ή τι θα παρακολουθούν καλύτερα οι δορυφόροι. Αυτό θα με ενδιαφέρει να μου το εξηγήσετε. Ευχαριστώ κύριο Σάγκνιου. Καλησπέρα Επίτροπε. Εγώ θα μιλούσω για τις αρρώσιμες καλλιέργειες και την απαγόρευση της λιφωσάτης. Λοιπόν, κοιτάξτε, θα πρέπει να το είδατε. Σας βλέπω να χαμογελάτε, αλλά είναι το χαμόγελο του δολοφόνου που έχετε για αυτό το θέμα που συζητάμε. Αυτό θα έλεγα εγώ. Οι Καναδοί πέρασαν ένα τεράστιο, τεράστια περίοδο δοκιμών για αυτή την ουσία και την περασμένη εβδομάδα στις Βρυξέλλες. Ήταν η συνεδρίαση της αντιγλυφωσάτης. Ακούστηκαν διάφορες λέξεις ορολογίας κλπ και αν βάλεις ε, μουστάρδα, δώσεις στα ποντίκια μουστάρδα ή αλάτι ή πιπέρι θα, θα πεθάνουν. Εμείς θέλουμε να μάθουμε τι γίνεται στην πραγματικότητα, στους κάμπους. Αυτό το υλικό επί 40 χρόνια το χρησιμοποιούμε. Δεν βρήκαμε να υπάρχουν παράστητα που αντιστέκονται, δεν κατάρρευσαν τα εδάφη μας, η απόδοση διπλασίασε μετά την ε, χρήση της λιφωσάτης. Και το άλλο που λησμονούν είναι η πλευρά της ασφαλείας των τροφίμων δεν πεθαίνουμε σαν τις μύγες μετά από 40 χρόνια που έχουμε εκτεθεί σε αυτή την ουσία ε, και υπάρχουν και εκείνοι που σαν και εμένα που είμαστε σαν τα καναρίνια στο ρηχείο που τουλάχιστον για 20 χρόνια έχουμε μου σκέψει, έχουμε σκεπαστεί από αυτή την ουσία θα έπρεπε να είμαι εδώ αν ήταν μεγάλο το πρόβλημα, θα είχα ζήσει Λοιπόν, παρακαλώ να αντέξετε απέναντι σε αυτούς. Θέλετε να σταματήσουν τις καλλιέργειες. Με, μετά η απαγόρευση των οικοτενοειδών. Όχι, θέλουν να το σταματήσουν και σε ανθοφορούσε καλλιέργειε και, και σε μη ανθοφορούσε καλλιέργειε. Τι θα κάνουμε ανταυτού. Ε, και θα είναι ό,τι κάνουμε άλλο θα είναι χειρότερο το περιβάλλον. Θα ψεκάζουμε τα πάντα. Με άλλες ουσίες. Πυρερυθρίνε. Λοιπόν, αντέξτε και απέναντι σε αυτού. Εγώ ήμουν μόνο στην αίθουσα τότε που ήμουν έτοιμο να μιλήσω υπέρ των γεωργών. Τέλο, άκουσα διάφορου που μιλούσαν για παγετό. Όλοι υπογράψατε για τη μείωση τη αλλαγή του κλίματο και όλοι θα μειώσετε τι εκπομπέ μεθανίου και εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακο για να μειώσετε τα έργα του θερμοκηπίου που παγιδεύουν τη θερμοκρασία. Φαίνεται σαν να τα καταφέρατε τελικά, διότι ε, ήρθε ο πα... παγετό. Λοιπόν, μαζέψτε τα και φύγετε, γιατί κραυγάζετε και αλλάζετε ασκόπου. Σα ευχαριστώ. Ο κύριος Λαζό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, οι ποσοστώσεις της ζάχαρης ε, λήγουν λίγουν στις 30 Σεπτεμβρίου που έρχεται. Ποια είναι τα σχέδια να καταπολεμήσετε την ισορροπία της αγοράς. Υπάρχουν ε, μέτρα που προβλέπονται στην επόμενη μεταρρύθμιση της κοινή αγροτικής πολιτικής για να αποφευθεί αυτή η ισορροπία. Και τι έχετε ε, προβλέψει για να αποφευθεί μια κρίση όπως αυτή κατά το τέλος των ποσοστώσεων των γαλακτοκομικών προϊόντων. Στην προηγούμενη συνάντηση με την κυρία Άγγελα Μέρκελ, ο κύριος Τρόμπ είπε ότι θα ξαναξεκινήσουν οι συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση για μια συνθήκη συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών. Πού βρισκόμαστε όσον αφορά αυτό το εγχείρημα. Τέλος, η κυρία Μάλστρομ συνάντησε τον Υπουργό ε, Οικονομικών του Μεξικού για να συναυθεί μια συμφωνία ελευθερών συναλλαγών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και Μεξικού. Θα γίνει 26 με 30 Ιουνίου στο Μεξικό ένα συνάντηση και μετά θα ακολουθήσει μια. κάθε μήνα θα υπάρχει συνάντηση. Τι γίνεται στον αφορά αυτή η μελλοντική συμφωνία και τι ακριβώ, ποια θα είναι η εμβέλεια αυτή τη συμφωνία με το Μεξικό. Αυτά και ευχαριστώ. Είχαμε πολύ καιρό για να έχουμε τέτοια σφοδρή συζήτηση. Πολύ δύσκολο το έργο σας κύριε Επίτροπε. Έχετε το λόγο. Thank you very much, uh, Chairman. Um, Ευχαριστώ. Να πω καταρχήν ότι ό,τι επιτύχουμε θα είναι για το συμφέρον των αγροτών, της ασφάλειας των τροφίμων, της ποιότητας και οι αγρότες είναι εκείνοι που μπορούν να επιτύχουν αυτούς τους στόχους όπως και οι στόχοι της ε, ε, βιωσιμότητας και της απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές. Ξέρουμε τα τελευταία χρόνια υπάρχουν κάποια προβλήματα εις ό,τι αφορά την ε, αντοχή της αγοράς, τη διαχείριση κινδύνων την εφαρμογή των συμφωνιών του 2015 για το κλίμα, για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Υπάρχουν προβλήματα σε ό,τι αφορά την προσέλκυση νέων στον ε, γεωργικό τομέα, στον τομέα των τροφίμων και το έχω πει πολλές φορές. Τώρα είμαστε σε μια φάση όπου αρχίζουμε να αναπτύσσουμε την πολιτική μας για να λύσουμε ορισμένα από αυτά τα προβλήματα. Μην ξεχνάμε και την έκθεση Ανδριού για την αγροτική ανάπτυξη. Μπορούμε να κάνουμε περισσότερα και στον τομέα των τροφίμων. Τώρα, τα θεμέλια της ΚΑΠ είναι τρία. Οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά. Ε, το οικονομικό κομμάτι είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί έχει να κάνει με την επιβίωση των αγροτών αλλιώς δεν θα έχουμε, προβλήμα, δεν θα έχουμε γεωργία ούτε απασχόληση ε, βεβαίως ε, είναι πολύ σημαντικές και οι περιβαλλοντικές πτυχές θα έλεγα λοιπόν ότι και ε, το θέμα του προϋπολογισμού είναι πολύ σημαντικό θα συνεχίσουν υπάρχουν εισφορές από τα κράτη-μέλη στον προϋπολογισμό καλή τύχη σε αυτό θα υπάρχουν συμφωνίες εις ό,τι αφορά την έκθεση Μόντι για πρόσθετους πόρους ε, στον προϋπολογισμό, περιβαλλοντική φορολογία. Θα πρέπει να το δείτε και αυτό. Εγώ θεωρώ ότι θα υπάρξουν κάποιες περικοπές στον συνολικό προϋπολογισμό και θα πρέπει να μεγιστοποιήσουμε αυτά που μπορούμε να επιτύχουμε για την Γεωργία. Αν μπορείτε να μου δώσετε περισσότερες πληροφορίες από τα κράτη-μέλη ότι μπορούν να το δουν διαφορετικά, θα ήταν πάρα πολύ σωστό. Εγώ πάντως στηρίζομαι στο... και εκείνο από την αρχή ότι όσο περισσότερα χρήματα έχουμε, τόσο περισσότερα θα, θα κάνουμε. Το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη είναι ένα θέμα. Ε, είχαμε πει το 15-16 να σταματήσουμε ε, να ε, το έχουμε στην παρέμβαση για την αποθεματοποίηση. Πολλοί στον κλάδο ε, χρησιμοποιούν το, το, το, τις εξελίξεις για να συμπιέσουν τις τιμές. Και εμείς ε, επεξεργαζόμεθα προτάσεις και μάθαμε από την εμπειρία του 2009 όπου είχαμε υποσοστώσεις και είχαμε εκείνη την εποχή ε, μεγάλη ποσότητα στην αποθεματοποίηση για να ε, τα χρησιμοποιήσουμε και να μην συμβιεστούν οι τιμές σε βάρος των αγροτών. Ε, οι τιμές ήταν χαμηλές αλλά τώρα εργαζόμεθα και με τρίτες χώρες και αξιολογούνται διάφορα προγράμματα για να δούμε πώς μπορούμε να δούμε τον επόμενο χρόνο το πρόβλημα αυτό για να μην ε, είναι ε, πολύ χαμηλή η τιμή. Μιλήσατε για τους κανόνες του ανταγωνισμού επίσης. τώρα έχουμε το, νομοθεσία Omnibus ε, που υπέβαλε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή Άγκρη. Τώρα ε, είναι επιτάπητος και η Κομισιόν πρέπει να ασχοληθεί, θα πρέπει να διαμορφώσουμε θέση. Ήμουν στον Καναδά και της είπα το τελευταίο δεκαήμερο για να βοηθήσω με τις εξαγωγές και να ε, δούμε τι ακριβώς γίνεται γιατί ήταν αντιφατικές οι ειδήσει. Τις επόμενες ε, δύο εβδομάδες θα μπορέσει να αρχίσει τριμερής διάλογος και θα προετοιμαστώ για να απαντήσω σε όλα τα θέματα λαμβάνοντας ε, υπόψη όλες τις απόψεις και με την Επίτροπο για τον Ανταγωνισμό συνεργαζόμεθα για να λειτουργήσει η πρωτοβουλία για ε, την ε, ε, αλυσίδα των τροφίμων η Επίτροπος θα συνεργαστεί και εγώ θα υποβάλω προτάσεις για την εφοδιαστική τροφική αλυσίδα προτάσεις ούτως ώστε να κινηθούν τα πράγματα και να μην υπάρξει μακρά περίοδος ανάλυσης των επιπτώσεων που θα επηρεάσει την καλύτερη νομοθεσία. Σίγουρα όμως θα πρέπει να είναι σωστή νομοθεσία. Τώρα για την θελοντική ε, συνδεδεμένη στήριξη, όλα αυτά είναι θέματα που θα πρέπει να, μας, ε, να τα δούμε. Κύριε Νίκολσον, καταρχήν ενεργοποιήθηκε το άρθρο 15 ε, και πριν περιμέναμε να κινηθεί η κυρία Μέη. Ε, προηγουμένως δεν, δεν μπορείτε να περιμένετε από εμά να αναλάβουμε δράσεις. Ε, ενεργοποίησε το άθρο, ε, προκήρυξε βουλευτικές εκλογές ε, και αυτό ήταν απροσδόκητο και τώρα θα πρέπει να περιμένουμε. Καταλαβαίνω γιατί προκήρυξε εκλογές και νομίζω ότι αξιοποίησε την ευκαιρία που της δίνεται. Έχει όμως τη δυνατότητα να κάνει με ήπιο ή σκληρό τρόπο ορισμένα πράγματα. Μπορεί να έχετε εσείς περισσότερες πληροφορίες από μένα αλλά όταν πήγα ε, και ε, μαζί με τον κύριο Μπαρνιέ και στις διάφορες συναντήσεις που έκανα και στη Βρετανία και στην Ιρλανδία είδα ότι ο διαπραγματευτή, το ομόλογο, το άλλο μέρος των διαπραγματεύσεων ε, θέλουν, θέλει να βρει λύσεις ε, γιατί ε, το, το εμπόριο μεταξύ Βρετανίας και Ιρλανδίας είναι πολύ σημαντικό. Πολλοί που παρευρέθηκαν στις συναντήσεις υπέβαλαν προτάσεις. Αν το Ηνωμένο Βασίλειο παραμείνει στην Τελωνιακή Ένωση αυτό θα βοηθήσει. Δεν ξέρουμε όμως τι θα κάνει γιατί ακόμα δεν έχει συσταθεί η διαπραγματευτική ομάδα. Σε 4-5 εβδομάδες αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι να συνεργαστούμε. Είμαι έτοιμος ως Επίτροπος να ε, συνεννοηθώ ε, και με την ε, κυβέρνηση της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου και τη Βόρεια Ιρλανδία να δούμε πώς θα βρούμε ρεαλιστικές λύσεις που θα μετριάσει τη ζημία για την οικονομία της Βρετανίας και της Ιρλανδίας. Πρέπει όμως να περιμένουμε μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Είμαι όμως ικανοποιημένος από την ενημέρωση, στην ε, λεπτομέρεια ε, στην οποία προχώρησε ο κύριος Μπαρνιέ και ως Επίτροπος σε σχέση με τα διαπεριφερειακά διαφορετικά ταμεία ε, διαθέτει μεγάλη εμπειρία εκεί. Τώρα, για τα βιολογικά προϊόντα ε, έχετε μια ενημερωτική συνάντηση ακριβώς μετά με τον κύριο Χόισλινγκ θα, θα σας ενημερώσει για όλα τα θέματα εκείνος αλλά θα πρέπει να έχουμε αξιόπιστο σύστημα για τα βιολογικά θα πρέπει να υπάρχει μια ακαιρεότητα και όλοι εργαστήκαμε με υπομονή το τελευταίο, το τελευταίο διάστημα για εναρμόνιση των κανόνων για τους Ευρωπαίους αγρότες και, τους, ε, και τις εισαγωγές από τρίτες χώρες. Επιτέλους υπάρχει πρόοδος. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τους σκιώδες για την πρόσφατη συνεργασία επ' αυτών των θεμάτων. Γιατί όλοι αντιμετωπίσαμε πιέσεις λόγω των καθυστερήσεων. Ε, πάντως, επί Μαλτέζικης Προεδρίας θα συνεχίσουμε για να φτάσουμε, να καταλήξουμε κάπου. Ε, υπάρχει πρόοδος εδώ. Τώρα, εις ό,τι αφορά τις ε, αντιδράσεις, ε, όταν έχετε 320.000, ε, θα γίνει κάποια καμπάνια και από τις μη κυβερνητικέ και τους αγρότες. Αλλά εδώ δεν είναι ποσοτικό το θέμα, είναι ποιοτικό. υπάρχουν και πολύ καλές παρεμβάσεις και θα ακολουθήσουν κι άλλες και το κοινοβούλιο σε ατομική βάση μπορεί να θέλει να κάνει παρατηρήσεις όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία. Δεν έχουμε, ε, έχουμε μια προθεσμία, αλλά δεν τελειώνει η ιστορία εδώ. Θα συνεχίσουμε να δεχόμαστε καλές ιδέες μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Έτσι κινείται η πολιτική. Θα ήμουν ευτυχής αν συμμετείχατε στην συνάντηση της 7ης Ιουλίου ε, που θα ε, κάνουν διαβουλεύσεις οι εμπλεκόμενοι, θα δούμε πώς αντιδρούν, θα υπάρχει ευκαιρία να δούμε πώς σχολιάζουν αυτά που έχουν ήδη υποβληθεί. Τώρα, ο εξυγχρονισμός της ΚΑΠ πρέπει να λάβει υπόψη του τη συμφωνία του 2015 για το 10, τις ε, συμφωνίες για τη διατροφή το 2015, τις ε, βιώσιμους αναπτυξιακούς στόχους, αλλά και τα εργαλεία που υπάρχουν ή δεν υπάρχουν ανάλογα με την περίπτωση. Υπάρχουν τομείς όπου όλοι συμφωνούμε ότι χρειάζονται και άλλα εργαλεία ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν οι γεωργοί την αστάθεια το, της αγοράς και να προσαρμοστούν στα προβλήματα. Έχουμε ανοιχτό πνεύμα σε ό,τι αφορά τις λύσεις, τη διαχείριση κινδύνων, την αστάθεια και την αβεβαιότητα για τους αγρότες. Αυτό σημαίνει εξυγχρονισμός. Ε, βέβαια, η παρούσα πολιτική δεν θέλουμε να ταλαιπωρεί τους αγρότες και να τους σε ό,τι αφορά δηλαδή την καταβολή των ενισχύσεων κλπ. Δεν θα επιστρέψουμε στις ε, ποσοστώσεις ζάχαρης. Η απόφαση ελήφθη πριν από πολλά χρόνια και τελειώνουμε τον επόμενο Σεπτέμβριο. Η ρύθμιση της παραγωγής δεν θα είναι κομμάτι αυτού που θα κάνουμε. Για το γάλα, πολύ μίλησαν για, και ο κύριος Χόισλιν για το γάλα. Η αγορά γάλακτος είναι ένα παράδειγμα του που θα πρέπει να εξυγχρονίσουμε την ΚΑΠ. Χρειάζεται να δοθούν περισσότερες ευκαιρίες για να αντιδράσουν οι αγρότες, να αξιολογήσουμε αυτό που θα κάνουμε, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε πιο καλά και πιο γρήγορα. Ε, ε σε κάποια κράτη-μέλη ε, έχουμε αύξηση 40% της τιμής του γάλακτος και 10% σε άλλα κράτη-μέλη. Δηλαδή υπάρχει κάποια βελτίωση. Ε, σε ορισμένα κράτη-μέλη είναι υψηλή η συγκέντρωση της αγοράς και δεν αξιοποιείται πλήρως η βελτίωση αυτής τη τιμές. Η μέση λοιπόν τιμή του γάλακτος τον περασμένο το Μάιο ε, ήταν 27 cents ανά χιλιόγραμμο, τώρα είναι 33,4. Το... Ε, αυτή είναι η αύξηση μέσα σε ένα χρόνο. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι, τα θέματα δεν έχουν πλήρως επιληθεί, κάθε άλλο. Αλλιώς δεν θα συνεχίζαμε στην, στον εξυγχρονισμό. Με την εξαίρεση του αποκορυφωμένου σε σκόνη, οι τιμές είναι παρόμοιες με το πενταετή μέσο όρο και υπάρχει και αύξηση 35% στο βούτυρο. Γενικά για το εμπόριο που αναφέρατε, ε, τώρα ε, επικαιροποιούμε την ε, συμφωνία με το Μεξικό μετά από 25 χρόνια. Μας προσφέρει ευκαιρίες για κάποια προϊόντα όπου είμαστε επιθετικοί όπως τα γαλακτοκομικά προϊόντα και μπορούμε να αυξήσουμε τις συναλλαγές γιατί δεν είχαμε πολύ εμπόριο στο, στα, με τα γαλακτοκομικά. είχαμε μόνο με τα προκυπευτικά. Είναι μια ευκαιρία λοιπόν τώρα με το Μεξικό να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Και στο τέλος του έτους περιμένουμε να αξιολογήσουμε αν θα ε, έχουμε ε, παρκείς συμφωνίες ελευθέρων συναλλακών. Δεν ε, νομίζω ότι υπάρχει βάση για φήμες ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε πρόκειται να κάνουν διαπραγματεύσεις για ζώνη ελευθέρων συναλλακών. δεν μπορώ να σταματήσω τις φήμες, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα ε, αρχίσει διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείε, αν δεν δει τη γενικότερη άποψη που ε, έχει ε, για το εμπόριο. γιατί οι θέσεις που διαμορφώθηκαν και παρουσιάστηκαν τον Σεπτέμβρη δεν βρήκαν σύμφωνη την Ευρωπαϊκή Ένωση. τώρα για το γλυφοσέιτ, γλυφοσάτε, ε, κάποιοι θα έλεγαν ότι εσείς και το κόμμα σας είναι οι δολοφόνοι, αλλά θα ε, είμαστε κόσμοι ε, απόψε. Οι εταιρείε φαρμάκων και έχουν, αλλά και οι αρμόδιες αρχές για, τα φάρμακα έχουν κάνει έρευνες και έχουν αναλύσει το προϊόν. Βέβαια, εσείς ερμηνεύσατε το χαμογελό μου ως κακό αποτέλεσμα. Ε, ε, δεν θα σας διαψεύσω τώρα, ε, θα δώσω όμως απαντήσεις. Πάντως εγώ υποστηρίζω μία επιστημονική προσέγγιση και αν η ο οργανισμός υπεύθυνος για τις χημικές ουσίες αποφανθεί θα δούμε ενδεχομένως θα συμφωνήσουμε με βάση τα επιστημονικά αποτελέσματα. Θα δούμε και θα εξετάσουμε το θέμα και στο Σώμα των Επιτρόπων αύριο. Σας ευχαριστούμε κύριε Επιτρόπε. Αν και δεν έλαβαν όλοι οι συναδέλφοι εξαντλητικές απαντήσεις και πλήρες απαντήσεις σε ερωτήσεις τους, αλλά ελπίζω να τις συμπληρώσετε και γραπτός. 20 συνάδελφοι ζήτησαν το λόγο, ένα λεπτό ο καθένας. Ο κύριος Σάνι ο πρώτος παρακαλώ. Ο Σάνι. Uh, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Δεν θέλω να μπω στη συζήτηση περί γλυφοσάτης. Έχω ιδιαίτερη άποψη γι' αυτό. Όλα είναι επιβλαβή πάνω από ένα συγκεκριμένο ποσοστό. Σε κανονικά επίπεδα μπορούμε να ανοιχτούμε πολλά. Επίτροπε, ανήκω σε αυτούς που ενδιαφέρονται για περισσότερες λεπτομέρειες. Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα εργασιών του επόμενου έτους. των φορέων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι στον τομέα ευθυνών σας. Θα ήθελα να ακούσω πληροφορίες, αν έχετε την καλοσύνη, σχετικά με τις αλλαγές που προβλέπετε για τον επόμενο χρόνο όσον αφορά την αγροτική πολιτική. Ε, λαμβάνοντας και τη δήλωση του ΚΟΡΚ 2. Η Γεωργία αφορά βάρη, τόνους, χιλιόγραμμα κλπ. Αλλά θα ήθελα να λάβουμε υπόψη και τον κόσμο και τον, την έννοια των ευφυών χωριών. Μια ιδέα που προωθείται και αναπτύσσεται. Θα ήθελα να αναπτύσσετε αυτό. Ο κύριος Νέκοφ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, όσον αφορά τον αυθόδη πυρετό των χείρων, ε, αυτό είναι κάτι που έχει πλήξει τις βαλτικές χώρες και την Πολωνία αλλά έχουν πληγεί και άλλες περιοχές. Την πανόλη των χείρων, μάλλον, συγγνώμη. Ε, όπως είναι η Βουλγαρία και η Ρουμανία κλπ. Ανησυχούν οι κτηνοτρόφοι στη Βουλγαρία για τον αυτό πυρετό των χείρων. Και έπρεπε να σκοτώσουν χιλιάδες ε, χείρους. Να θανατώσουν χιλιάδες χείρους. Σε περιοχές ε, όπως είναι η Γκριμούντα που έχει μεγάλη κτηνοτροφία και παραγωγή χειρίου κρέατος. Έχουμε και ένα είδος χείρου από τα Ανατολικά Βαλκάνια που υποτίθεται ότι προστατεύεται σαν είδος. Και ανησυχούμε για αυτή την, ε, αυτό το είδος του χείρου σχετικά με την ασθένεια αυτή. Ε, Έκλεισε απευθύνω περισσότερο παρά ερώτηση. Σας παρακαλώ, μπορείτε να μας δώσετε κάποιες ιδέες, θα διατεθούν περισσότερα χρήματα, ούτως ώστε να καταπολεμηθεί αυτή η ασθένεια των χείρων. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Δεν χρειάζεται να σας πω, Επίτροπε, πόσο ζωτική σημασία θα είναι οι διαπραγματεύσει του Brexit για τη δημοκρατία της Ιρλανδίας. Και θα χαίρεστε που κάποιο από την Ιρλανδία είναι εδώ παρόν σήμερα. Θα πρέπει λοιπόν να δεχτούμε ότι υπάρχουν αντικρώμενα μηνύματα που εμφανίζονται για την πορεία των πραγμάτων. Απ' τη μία ακούμε ότι είχαμε επιτυχίες που όλοι πίστευαν θα έχουμε. Δηλαδή, αν καταλήξουμε με μια ενωμένη Ιρλανδία, οι έξι κομιτείε θα μπορέσουν να ενωθούν με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώ έλεγε ότι αυτό θα είναι πρόβλημα. Ευχαριστούμε που ήσασταν ένα πρόβλημα που ήταν ανύπαρκτο. Έχουμε όμω προβλήματα ενδεχομένω με την ελεύθερη διακίνηση αγαθών και ανθρώπων. Και έχουμε ένα πρόβλημα με τη στάση τη Ευρωπαϊκή Επίτροπή. Ακούμε κάποια πράγματα, Όπω, δεν θα δώσω παραπάνω από 30 λεπτά την εβδομάδα. Το Brexit ποτέ δεν θα είναι επιτυχέ. Ο Γκίβερ Χόφστατ πριν τον Brexit είπε ότι η Βρετανία θα είναι πολιτικός νάνος. Ανησυχείτε. Και θα ήταν δικαιολογημένο να ανησυχούσατε. Ανησυχείτε ότι οι διαπραγματεύσει θα βασιστούν στο πείσμα και, το, και Είναι σαν να χωρίζει ένα ανδρόγυνο. Σαν να πενδιαζύγει ένα ανδρόγυνο. Λοιπόν, η εξαγωγή και η εισαγωγή τη Βρετανία και τη Ιρλανδία και τη Ολλανδία θα είναι τα θύματα. Και αυτοί που εργάζονται για την BMW για την BMW στη Γερμανία. Πιστεύετε ότι θα, θα, θα ξοδέψουν, θα χρησιμοποιήσουν πάνω από μισή ώρα την εβδομάδα για τι διαπραγματεύσει. Εσεί θα αφιερώνετε παραπάνω από μισή ώρα την εβδομάδα για τι διαπραγματεύσει. Ξέρετε πόσο ζωτική σημασία είναι. Ο κύριο Δεκάστρο, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ ε, κύριε Επίτροπε που είσαστε παρόν. Ευχαριστούμε που υπενθυμίσατε ότι αυτή η Επιτροπή στη συνεδρίαση στις 3 Μαΐου που πέρασε ε, ενέκρινε τον κανονισμό Omnibus. Ήταν η πρόταση κανονισμού μας ε, στο χρόνο που είχαμε καθορίσει. Η Επιτροπή Προπολογισμών είχε αναπέψει ε, το θέμα στις 20 Μαΐου. Κοιτάξτε τώρα, έχω μια ερώτηση πολύ απλή. Ξέρετε και όπως υπενθυμίστηκε ότι έχουμε ξεπεράσει τον κανονισμό Omnibus. Κάναμε περισσότερα πράγματα. Κάναμε προτάσεις προς όφελος της Γεωργίας προσπαθώντας να δώσουμε μια απάντηση στα μεγάλα προβλήματα που αφορούν την εσωτερική αγορά, τη διαχείριση των κινδύνων. Εκμεταλλευόμενοι την πρότασή σα, ξεπεράσαμε τα αρχικά όρια. Η ερώτησή μου είναι απλούστατη. Το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, οι Υπουργοί τη Γεωργία ενέκριναν μια γνωμοδότηση επί Μαλτέζικη Προεδρία που ουσιαστικά δεν λέει τίποτα ή σχεδόν τίποτα. Αυτή η θέση περιορίζεται μάλλον κάνει επαναχωρήσει και στην ε, αρχική πρόταση, πρόταση. Λοιπόν, στου τριμερεί διαλόγου, αυτή είναι η ερώτησή μου, στου τριμερεί διαλόγου. Όπω το έθεσε και ο συνάδελφο Άντριο. θα έχουμε σύμμαχο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτω ώστε να κινηθεί το Συμβούλιο προ κάποιε δικέ μα ενδείξει και κατευθύνσει ή αντίθετα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, κατευθύνεται προ μια νέα νομοθετική πράξη που ίσω κατά τη διάρκεια αυτή τη ε, θητεία θα είναι δυνατόν να περάσει και να θεσπιστεί. Η κυρία Εράνς Καρσία. Ευχαριστώ. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον Επίτροπο γιατί αν κατάλαβα καλά, επιτέλου θα καταθέσω την πρόταση για την τροφική αλυσίδα, που την περιμένουμε πω και πώ εδώ και πολύ καιρό, γιατί έχει καθυστερήσει. Χαίρομαι πάντως που επιτέλου θα το κάνετε. Επίση, ε, είπατε ότι σίγουρα θα έχετε το χρόνο για πραγματική μεταρρύθμιση τη κοινή γεωρικής πολιτική. Αυτό με εξέπληξε, γιατί αν παίρνουμε ε, αν περιμένετε την ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν ξέρω αν θα έχετε αρκετό χρόνο. Λάβατε υπόψη κατά την εξέταση του Brexit και του δημοσιονομικού του όρου την ύπαρξη της Βρετανικής επιταγής. Τι κονδύλια θα απαιτήσει από τον κυρωτικό προπολογισμό και μάλιστα ετησίω, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον πρωτογενή τομέα και ιδιαίτερα για τον πρώτο πυλώνα της κοινή γεωργικής πολιτικής. Ευχαριστώ. Κύριο Στάκουλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν συμφωνείτε μαζί μου ότι η κοινή γεωρική πολιτική θα πρέπει να εξασφαλίζει τη συνέχιση της παραγωγής σε όλους τους τομείς, ακόμη και στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές, τις περιοχές που αντιμετωπίζουν κάποια μειονεκτήματα. Πιστεύετε ότι θα καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε μια βιωσιμότητα της παραγωγής ακόμη και στις πιο μειονεκτικές περιοχές μετά τις προτάσεις, τις τελευταίες. Επίσης, είναι δυνατόν ε, να, κρατήσουμε τα βιολογικά χαρακτηριστικά μιας παραγωγής όταν δεν υπάρχει αυτή η συνέχεια. Εγώ θα ήθελα να υπάρχει τέτοια συνέχεια γιατί οι τοπικοί πληθυσμοί εξαρτώνται από αυτό και νομίζω ότι αν σταματήσει η εξαίρεση για τα οριθετημένα παρτέρια θα είναι πολύ δύσκολο για τους δικούς μας παραγωγούς να συνεχίσουν τη βιολογική παραγωγή. Ξέρετε ότι έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη σε εσά και περιμένουμε πολλά από εσά. Δεν θα πρέπει να μείνετε στην ιστορία ως ο επίτροπος που οδήγησε σε αφανισμό τη βιολογική παραγωγή στις σκανδιναβικές περιοχές και χώρες. Ευχαριστώ κύριε Νόιχλ. Και εγώ έστειλα ερωτήσεις προς ε, ε, εσάς και καλό είναι να τις επαναλάβω. Θα ε, ήθελα να επαναλάβετε αυτό που είπατε ότι πρέπει να βρούμε και άλλες αγορές. ερωτώ και έχω στείλει σχετική επιστολή αν δεν έχετε αλλάξει άποψη στην Κομισιόν ε, ό,τι αφορά την ε, διεύρυνση της παραγωγής. Δηλαδή δεν θα πρέπει να έχουμε εξωτερικό εμπόριο συν ε, ενώ όλοι οι άλλοι θα έχουν αρνητικό πρόσημο. Συγκεκριμένα και μου έκανε ε, ε, προηγουμένως και αυτό με εξέπληξε, περιγράψατε θετικά την εξέλιξη για το οργανισμό Omnibus. Ε, νομίζω ότι ε, προσπαθείτε να περάσετε σε μια νέα εξελιγμένη ΚΑΤ. Η τροποποίηση από την πίσω πόρτα γίνεται ε, εν προκειμένου στην ΚΑΤ όμως δεν ήταν αυτό το πνεύμα των διαπραγματεύσεων για το Όμνιμπους. Ε, υπήρξε ε, ε, κάποια, ε, κάποια βελτίωση θα έπρεπε να γίνει στο, στην ΚΑΠ, αλλά δεν νομίζω ότι θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με γενικότητες και χωρίς να διαφοροποιείτε τα θέματα. Ε, από τη μία ε, θέλετε να ε, προβλέψετε διάλογο και από την άλλη βιάζεστε χωρίς διαβουλεύσεις με τους ειδικού να λάβετε τις αποφάσεις σας. Και αυτό το βρίσκω άκρος αρνητικό. Ναι, αυτή είναι μια γενική ερώτηση. Αν δηλαδή ο κανονισμός Omnibus πρέπει να επισέρχεται και σε θέματα που κανονικά ανήκουν στο μέλλον της ε, κοινή γεωρικής πολιτικής. Ή μήπως θα πρέπει από τώρα πιλωτικά να ελέγξουμε κάποιες δράσεις στα πλαίσια των αλλαγών, ώστε αργότερα μετά το 2006 και αφού το έχουμε δοκιμάσει και πιλωτικά κάποια θέματα να μπορέσουμε να τα εφαρμόσουμε. Ο κύριος Δενανό. Ευχαριστώ κύριε Επιτροπέ. Έχω, είχα να θέσω μια ερώτηση για τον Brexit, αλλά μια και τον ανέφεραν πολλοί άλλοι συνάδελφοι, δεν θα σταθώ κι εγώ σε αυτό. Έχω κάποιες ερωτήσεις για το πρόγραμμα Leader, που είναι πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Και ως πρώην Περιφερειάρχης ε, έχω πολλές προσδοκίες από το πρόγραμμα Leader και θέλω να διατηρηθεί και κυρίως να απλουστευτεί, γιατί υπάρχει πρόβλημα στην εφαρμογή του και πολλές καθυστερήσεις στα τελευταία προγράμματα, leader. Δεύτερη ερώτηση αφορά τη ζάχαρη και την κατάργηση των ποσοστώσεων ζαχάριος. Δεν θεωρείτε ότι αυτή η κατάργηση των ποσοστώσεων ίσως ε, έρθει σε αντιπαράθεση με την αναθεώρηση της οδηγίας για την ενέργεια και ιδιαίτερα για τα βιοκαύσιμα πρώτης γενιάς ε, που θα η χρήση των οποίων θα πρέπει να μειωθεί ε, σε ό,τι αφορά τα καύσιμα αυτοκίνη για τα οχήματα. κυρία Πετήρ και εγώ ασχολούμαστε με το θέμα αυτό και εκεί πραγματικά προβληματιζόμαστε μήπως ε, η μείωση των βιοκαυσίμων πρώτης γενιάς επηρεαστεί από αυτή την κατάργηση των ποσοστώσεων στη ζάχαρη. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Καπούτο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, κύριε Χόγκαν που ήρθατε. Δεν θα επαναλάβω τις τεθείς ερωτήσεις, θα μπω συγκεκριμένο για την ξυλέλα. Η απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν έχει τροποποιηθεί κατόπιν των ετοιμάτων της περιοχής της Πούλια, ξεκινώντας από το άρθρο 5 που επιτρέπει να ξαναφυτευτούν φυτά στην περιοχή που έχει πληγεί. Σύμφωνα με εκτίμηση που έγινε στην περιοχή, οι ζημιές είναι περίπου του ύψου ενός δισεκατομμυρίου ευρώ από αυτό. Ερώτηση, θα επιστραφούν αυτά τα χρήματα, θα αποζημιωθούν οι γεωργοί που επλήγησαν από αυτή την ασθένεια, τα φυτά τους. Όσον αφορά τα ελαιόδεντρα που, έχουν, που είναι στις περιοχές αυτές. Η Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΤΕ τέλος του Μαρτίου έδειξε ε, ε, πρόθυμη να βοηθήσει να, γίνουν, να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. Τώρα όμως διστάζει. Θα εφαρμοστεί η ληφθής απόφαση. Τι προτίθεστε να κάνετε. Κατά κάποιο τρόπο θα προβλεφθεί μια κάποια στήριξη, μια αποζημίωση για όλους ε, τους ε, ελαιοκαλλιεργητές που έχουν πληγεί από το πρόβλημα της ξυλέλα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Η κοινή αγροτική πολιτική ε, προσαρμόζεται στην πραγματικότητα. Η χρηματοδότηση όμως και αυτή μεταβάλλεται. Σε αυτές τις περιστάσεις Πώς μπορείτε να στηρίξετε τα κράτη-μέλη εκείνα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά τη χρήση των σωστών οικονομικών μέσων για τη στήριξη των μικρών εκμεταλλεύσεων, διότι αυτοί οι δικαιούχοι αντιμετωπίζουν αυξανόμενες δυσκολίες για την εξασφάλιση συγχρηματοδοτήσεως προγραμμάτων και όσον αφορά την επένδυση των καταλήλων ποσών για να υλοποιηθούν τα προγράμματά τους. Μια άλλη ερώτηση με την απόσυρση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και με την απώλεια της συμμετοχής της χώρας αυτής στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Το αναφέρατε κι εσείς άλλωστε αυτό. Ένα πολύ σημαντικό ποσό θα χαθεί και θα μειωθεί το κονδύλι για την ΚΑΠ. Λοιπόν, ποια είναι η δυνατότητα να πετύχουμε τους στόχους σύγκλησης ε, με τη χρήση του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, λαμβάνοντα αυτά υπόψη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Επίτροπε. Μια σύντομη ερώτηση έχω για τα θέματα, τα βιολογικά, για τις βιολογικές καλλιέργειες. Εξέφρασα ανησυχίες όταν παρουσιάστηκε η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αυξήθησαν ε, οι ανησυχίες μου. Υπάρχουν πολλές ανησυχίες στους βιολογικούς καλλιεργητές στην Ευρώπη. Ποια θα είναι η κατάσταση στο μέλλον, το προτινόμενα μέτρα πότε θα υθετηθούν. Συζητείτε εκτενώς επιμακρών. Στις 11 Μαΐου συνέβη κάτι εξαιρετικό στη Σουηδία. Η, η Προεδρία του Οργανισμού για την Προστασία της Φύσης στη Σουηδία, η Ένωση Βιολογικών Παραγωγών, ο Πρόεδρος Ενώσεως Γεωργών, ο Πρόεδρος της Ενώσεως βιολογικών καλλιεργητών, καλλιεργητών βιολογικών προϊόντων και ο πρόεδρος προστασίας καταναλωτών έκανε κοινή ανακοίνωση τύπου. Είπαν ότι ανησυχούν πάρα πολύ για τα αποτελέσματα όσον αφορά την παραγωγή βιολογικών προϊόντων πληρώνονται για αυτά που παράγουν. Αμείβονται καλά στη Σουηδία οι καλλιεργητέ βιολογικών προϊόντων, διότι και οι καταναλωτέ είναι έτοιμοι να καταβάλουν το τίμημα. Αν περάσει αυτή η πρόταση, κυρίω όσον αφορά τι καλλιέργειε στο βορρά, θα καταστραφεί η αγορά. Στη δυτική Σουηδία έχουμε ακόμα 0 βαθμού. Ακόμα περιμένουμε την πρώτη εβδομάδα που θα ανέβει πάνω από το 0 θερμοκρασία και προσπαθούν να μας υποχρεώσουν να πάψουμε να καλλιεργούμε. Τίποτα δεν έχει αναπτυχθεί ακόμα, διότι ε, είναι, δεν μπορούν να βγουν τα φυτά γιατί είναι παγωμένη η ατμόσφαιρα. Είχα ακόμα την περασμένη εβδομάδα υπό το μηδέν. Τι έχετε να πείτε έναντι αυτών των εκπροσώπων των διαφόρων, των διαφόρων συμφερόντων που ανέφεραν σε αυτές τις ανησυχίες των ανακοινωθέν τους για τον τομέα. Ε, δεν έχετε μόνο Σουηδία κρύο. Ο κύριος Ντόρφμαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, και θέλω να αναφερθώ και εγώ στις επιφυλάξεις ε, κάποιων συναδέλφων σε σχέση με τα, την online συζήτηση. Ελπίζω να γίνει σωστή ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Είναι κρίμα όμως ε, για τη διάσκεψη το, στις Βρυξέλλες ε, δεν λήφθη υπόψη το Κοινοβούλιο γιατί συμπίπτει με τη σύνοδό μας την ε, μηνία. Ε, θα θέλαμε να συμμετάσχουμε καλύτερα. Τώρα δύο πράγματα. Η κυρία Μούλερ μίλησε για τους όψιμους παγετούς. Ήταν μεγάλο το πρόβλημα και είναι ακόμα στην Ευρώπη. Υπάρχουν μεγάλες περιοχές που επλήγησαν και η ζημία ήταν πολύ μεγάλη ε, ορισμένε φορές. Ε, ε, έγιναν ε, φαντάζομαι συζητήσεις για παρέμβαση. Ένα άλλο θέμα που συζητείται στη Γερμανία είναι ο ρόλος και η επιστροφή των αρπακτικών του λύκου που έχει πάρει απειλητικές διαστάσεις στην γεωργία, στην παραδοσιακή γεωργία μικρά ζώα ε, αντιμετωπίζουν μεγάλους κινδύνους. Ε, ίσως λοιπόν θα έπρεπε να υπάρχει ρύθμιση ε, αυτών των αρπακτικών ζώων λύκου, αρκούδας στα κτηνοτροφικά ζώα. Ίσως θα έπρεπε να το δούμε αυτό και να φροντίσουμε να... Ε, επίσης πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ γεωργίας και προστασίας της φύσης ε, που δεν υπάρχει θεωρώ γιατί η ισορροπία πηγαίνει υπέρ της ε, προστασίας της φύσης προβολικά. Ευχαριστώ κύριε Χόιμπουχ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Επίτροπε, δεν μπόρεσα να παρευρεθώ σε όλη τη συνεδρίαση. Έπρεπε να πάω στην Ολομέλεια και δεν ξέρω αν ε, θίξατε το θέμα. Αλλά στις γραπτές ερωτήσεις, στα πλαίσια του διαφορετικού ε, διαλόγου, θέσαμε ερωτήσεις για τη συγκέντρωση της γεωργίας. Δεν συμφωνώ με την, ε, τις απαντήσεις απόλυτα, πρέπει να πω. διότι η θεωρείται υπεύθυνη τη Γενική Διεύθυνση για την Εσωτερική Αγορά. Σίγουρα η Γενική Διεύθυνση έχει ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Ε, τα, ε, ε, τα κράτη-μέλη τα κάλεσε να παρουσιάσουν απαντήσεις για τις συστάσεις, αλλά δεν είχε ολοκληρωθεί το θέμα, ούτε είχαν γίνει επισκέψεις επιτόπου. Ε, είναι πολύ σημαντικό να δούμε τη βάση της ε, γεωργίας. Ε, δεν μπορούμε δηλαδή να στέλνουμε, να, θεωρούμε ότι υπεύθυνοι είναι κάποιοι άλλοι που δεν είναι στον τομέα της γεωργίας. Θα πρέπει να δούμε επίσης τι συνέχεια θα δοθεί ε, στην έκθεση του Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία σχετικά με τη συγκέντρωση στη Γεωργία. Υπάρχουν κάποιες ε, κατευθυντήριες γραμμές ε, εθελοντικές. Πώς θα πραγματοποιηθούν, δεν μπορεί να είναι υπεύθυνη μόνο η Γενική Διεύθυνσή για το θέμα αυτό. Ε, υπάρχουν επίσης ορισμένες δομές εταιριών holding που επίσης θα πρέπει να μας απασχολήσουν. στο διάλογο από πέρα. ο κύριος Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και για τη σωστή προφορά του επιθέτου μου. Είχα στείλει στον Επίτροπο μία ερώτηση για τον κανονισμό Omnibus και τη δυνατότητα ορισμού της έννοιας της ε, ενεργού καλλιέργειας. Στη Φλάνδρα ο ορισμός αυτός είναι που δίνει ενάυσματα στους ε, νεαρούς γεωργούς για να συνεχίσουν την οικογενειακή γεωργική εκμετάλλευση ε, παρά τις τεράστιες πιέσεις που ασκούνται σε επίπεδο τιμών. Βέβαια, είπατε ότι και εσείς προβληματίζετε και σε ενδιαφέρει ε, το μέλλον των νέων Γιώργων και χαίρομαι γι' αυτό και αν όντως ε, προβληματίζεστε να το αποδείξετε εμπράκτος. Πώς από τη μια λέτε σας ενδιαφέρει το μέλλον των νέων και από την άλλη περιορίζετε σημαντικές ε, ευκαιρίες για αυτούς. Επίσης υπάρχει dumping σε ό,τι αφορά τους μεταποιητές για ομίλων. Έγινε κάποια έρευνα την οποία είπατε ότι γνωρίζετε και υποσχεθήκατε ότι σε ένα μεταγενέστερο στάδιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προσφέρει νομική βοήθεια στη, στους ε, παραγωγούς γεωμήλων. Σε τι φάση βρίσκεται αυτή η αντιδικία με τη Βραζιλία για το θέμα αυτό. Ε, κυρία Ριμπέιρο, κύριε Επιτροπέ, πριν από δύο εβδομάδες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε την πρόταση για την ε, διεύρυνση του πεδίου εφαρμογή του άρθρου 349 τη Συνθήκη για τη Λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να ισχύσουν κάποιες ειδικέ εξαιρέσει για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές σε πολλούς κανονισμούς και όχι μόνο στον κανονισμό ΠΟΣΕΙ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω τι γίνεται με τις δύο προτάσεις ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η πρώτη αφορούσε την ε, εκ των προτέρων ε, μελέτη επιπτώσεων των εμπορικών συμφωνιών στις εξ, εξόχως απόκεντρες περιοχές. Δεύτερη πρόταση που κάναμε είναι να προταθούν διαφοροποιημένα μέτρα και εξαίρεση σε περίπτωση που υπάρχουν κρίσεις αγοράς για τις ε, εξόχως απόκεντρες περιοχές, ώστε οι ενισχύσεις ε, που θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα κράτη-μέλη να προσαυξάνονται οι ενισχύσει αυτές για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές ε, προκειμένου να στηρίξουμε τους γεωργούς αυτών των περιοχών. Ποια είναι η θέση σας απέναντι στις δύο αυτές προτάσεις που συγκεκριμένα υποβάλαμε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γιάρ. Äh, Ευχαριστώ πολύ. Τρεις σύντομες συμπληρωματικές ερωτήσεις. Πρώτον, οι online διαβουλεύσεις Μπορούμε να το δούμε με διαφορετικού τρόπου το θέμα. Μένα δεν μου αρέσει να συμμετέχουν μόνο πέντε χώρε μέλη. Παρακαλώ τον ε, Επίτροπο να φροντίσει να γίνονται διαβουλεύσει όπου θα συμμετέχουν και 28. Τώρα για τη διαδικασία Omnibus είχαμε σίγουρα εξαιρετικέ ε, ιδέες που τις ε, εγκρίναμε εδώ για την αγροτική μεταρρύθμιση είχαμε πει ότι θα ξεπεράσουμε το 2020, θα δίναμε χρόνο δηλαδή για να γίνει μια εκτενή συζήτηση για την επόμενη μεταρρύθμιση. Δεν ξέρω εσείς προσωπικά τι πιστεύετε γι' αυτό. Για τις κατεξουσιοδότηση πράξης στην Γερμανία ακούσαμε στο ροδιόφωνο ότι ε, ε, δεν ε, ε, έχουμε, έχουμε αρχίσει να έχουμε προβλήματα ε, λόγω των αλλαγών στην καλλιέργεια λευκοματούχων φυτών και σόγιας. δεν ξέρω δηλαδή αν έχετε πρόγραμμα διαφοροποίησης στην καλλιέργεια αυτών των φυτών. Και τέλος τα βιοκαύσιμα πρώτης γενιάς, τα αυτά, τα βιοκαύσιμα πρώτης γενιάς θα πρέπει να ε, φροντίσετε να μην, να μην ε, αντιμετωπιστούν με τέτοιο τρόπο ώστε να υπονομεύσουν τις προσπάθειες για το κλίμα. Ο κύριος Μπούντα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον Επίτροπο που ήρθε για αυτό το διαρθρωμένο διάλογο. Θα ήθελα να σας ενημερώσω για μία ε, βόλτα που έκανα τις προάλλες στις Βρυξέλλες. Στον ελεύθερο μου χρόνο προσπαθώ να έρθω σε επαφή με γεωργούς ε, στο Βέλιο και μάλιστα πηγαίνω απροειδοποίητος για έκπληξη ε, για να δω την πραγματική κατάσταση και ε, βρήκα μια γεωργική εκμετάλλευση που κατάφερε να αντισταθεί στην κρίση της αγοράς γιατί έχουν μηχανισμούς για τη διάθεση των προϊόντων τους με το δικό τους κατάστημα και τους δικούς τους πελάτες. Βέβαια, γύρω από την γεωργική αυτή εκμετάλλευση, πολλά εκτάρια προσπόληση, γιατί οι γειτονικοί γεωργοί δεν είχαν αντίστοιχου μηχανισμού για να ανταπεξέλθουν στι προκλήσει αγορά. Μετά πήγα σε μια άλλη γεωργική εκμετάλλευση, ε, γαλακτοκομική μονάδα, που τη διαχειρίζονταν δύο νεαροί γεωργοί, ε, που μου είπαν ότι σε, σε 12 χρόνια μόνο δύο φορές ε, πήγαν διακοπές μου είπε ο ένας από τους δύο, ενώ ο άλλος μου είπε ότι είναι τεράστια η γραφειοκρατία. Είχαν 80 κεφάλια, αλλά παρόλα αυτά τα βρήκα σκούρα με τη γραφειοκρατία, γιατί δεν έχουν προσωπικό και το μισό τους προσωπικό προσπαθεί να ανταποκριθεί στις γραφειοκρατικές διατυπώσεις. Και στη Ρουμανία ένας Γιώργος πρέπει να συμπληρώσει 45 σελίδες Έτηση για να έχει πρόσβαση στις ευρωπαϊκές ενισχύσεις, στις γεωργικές ενισχύσεις. Και όταν μιλήσουμε για ενισχύσεις για βόλιο και χείριο κρέας, ε, χρειάζεται να περάσει πολλούς χρόνους μέχρι να υποβάλει τα χαρτιά του Γιώργος για να μπορέσει να λάβει ενίσχυση. Ευχαριστώ πολύ, Επίτροπε. Η ερώτηση αφορά ε, τα αυγά από κότες ελεύθερης βοσκής. Έχουν υποφέρει οι εκμεταλλεύσεις όταν έχασαν το καθεστώς ελεύθερης βοσκής μετά τη χρηματοδότηση. Όταν είχαμε ε, το, τη γρήπη των ε, πτηνών, ε, θέλαμε να βρούμε μια λύση μέσω κατάλληλης νομοθεσίας. Δεν υπήρξε καιρός να κινηθούμε κατάλληλα. Τώρα, μετά αυτή την επιζωοτία για να μην ξανασυμβεί αυτό. Πώς μπορούμε να βρούμε μια λύση. Δεύτερον, υπάρχουν δυνατότητες χρηματοδότησης για να καλυφθούν οι απώλειες των ε, γεωργών. Ποιες είναι οι απαιτήσει και οι προϋποθέσεις. Υπήρξε ενδιαφέρον στην Ολλανδία. Οι ίδιοι οι γεωργοί θέλουν να συλλέξουν κάποια χρήματα. Και με αυτά τα χρήματα ίσως να πετύχουν κάποια συγχρηματοδότηση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Επόμενος. Πετήρ. Η ε, κυρία Πετήρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε. Σας ευχαριστώ που το Μάρτιο ήρθατε στο Ζάγκρεπ για ένα σχέδιο στο οποίο είμαι εγώ πρέσβυρα του καλύτερου νεαρού γεωργού γιατί έτσι προωθούμε ε, ευρηματικά, βιώσιμα και καινοτόμα σχέδια γεωργίας. Βλέπουμε δυστυχώς πολλούς νέους να εγκαταλείπουν την Κροατία αναζητώντας ε, μία απασχόληση και μάλιστα το τελευταίο χρόνο 80.000 ε, συμπολίτες μου εγκατέλειψαν την πατρίδα τους αναζητώντας μία καλύτερη δουλειά. Και δυστυχώς ε, φεύγουν ενώ στις, ε, στην πατρίδα τους υπάρχει δυναμικό, ιδιαίτερα στη Γεωργία υπάρχει ε, δυναμικό προς αξιοποίηση. Φαίνεται ότι δεν, τους, δεν είναι αρκετά δελαστική για αυτούς η Γεωργία ή φοβούνται ότι αν ασχοληθούν με τη Γεωργία η παραγωγή τους δεν θα βρει διέξοδο λόγω των αθέμητων εμπορικών πρακτικών. Βέβαια η, Κροατία έχει κάποιο ηθικό μηχανισμό για την προστασία από τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές, αλλά δεν αρκεί αυτός ο εθνικός μηχανισμός. Ερωτώ λοιπόν, σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, θα πρόκειται να θεσπίσετε κάποια μέτρα προκειμένου να μπορέσουν οι γεωργοί να έχουν κάποιες πιο βιώσιμες γεωργικές δραστηριότητες, οι νεαροί γεωργοί κυρίως, ο κύριος Σέκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επίτροπε Χόγκαν, ε, για λόγους σεβασμούς για το υψηλό σας αξίωμα δεν θα ε, κάνω σκληρή κριτική ούτε θα κάνω δολοφονικά χαμόγελα. Για το μέλλον της ΚΑΠ όμως πιστεύω ότι χρειάζεται να υποβάλλετε καλύτερες προτάσεις για να αντιμετωπίσετε την ανάγκη διατήρησης της υγείας ανθρώπων, ζώων, τη βιοπικιλότητα και να επιτύχετε και τους κλιματικούς στόχους. Για την επίτευξη της ε, Συμφωνίας των Παρισίων είναι πολύ σημαντικό η παραγωγή κρέατος και γαλακτοκομικών να μειωθεί ούτω ώστε να μειωθούν και ε, οι ε, σχετικές βλαβερές εκπομπές. Πώς βλέπετε να γίνεται αυτό ε, διατηρώντας την ανταγωνιστικότητα. Εμείς τώρα έχουμε μια υπερπαραγωγή, πολύ μικρή παραγωγή ε, καταστράφηκαν και εντατικοποιείται η γεωργία συνεχώς. Η ανταγωνιστικότητα λοιπόν εξελίσσεται αρνητικά πιστεύω εγώ και οι επιπτώσεις αυτού του μοντέλου αφορούν και χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου καταστρέφουμε τοπικές αγορές στην Αφρική και σε άλλες χώρες και δημιουργούμε προϋποθέσεις φυγής από εκεί. Η ανταγωνιστικότητα πάντοτε ε, αποβαίνει σε βάρος της ποιότητας, της βιοπικιλότητας κλπ. Είναι πάρα πολύ ψηλό το τίμημα. Ο Επίτροπος ε, τι γνώμη έχει για το ζήτημα αυτό. Ευχαριστώ. Μαγκίνες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Μ' αρέσει ο διαθρωμένο διάλογο, αλλά μακάλα μην γινόταν το βράδυ, γιατί το Προεδρείο του Κοινοβουλίου συνεδριάζει το βράδυ της Δευτέρα, Ζητώ συγγνώμη την Επιτροπή που απουσιαζάει. Βοηθό μου με ενημέρωνα για τα θέματα και τι απαντήσει Ευπρόσθετα τα σχόλιά σα για, ε, για το φοδιασμό σε τρόφιμα και την αλυσίδα των τροφίμων. Θα συνεργαστούμε μαζί σα, πάνω σε αυτό, Επίτροπε. Δεύτερον, όσον αφορά τα σχόλιά σα για το Brexit, η Ιρλανδία, το κάτω μέλο μου, θα πληγεί περισσότερο. Οι συνάδελφοι στην αίθουσα γνωρίζουν ότι αν υπάρξει πρόβλημα όσον αφορά το βόλιο κρέα τη Ιρλανδία ή το κομικό τομέα λόγω κακή συμφωνία του Brexit, θα επηρεαστεί και η αγορά τροφίμων τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Νομίζω ότι έχουμε υποστήριξη σε αυτή την αίθουσα. Και η επίσκεψη του Μισελ Μπαρνιέ στα σύνορα την Παρασκευή ήταν ενημερωτική. Διότι υπήρχαν κάποιοι εκπρόσωποι του τομέα που ανέφεραν κάποιε λύσει και αυτό θα πρέπει να δούμε και ελπίζω να μπορέσουμε να συνεργαστούμε από αυτού συγκεκριμένο σημείο σχετικά με την κοινή εγωτική πολιτική. Γίνεται λόγος ε, για περιοχές που εστιάζονται ιδιαίτερα στον αφορά του οικολογικούς σκοπούς. Θα πρέπει να υπάρχει ποικιλομορφία και αμυψισφορά όσον αφορά τις καλλιέργειες. Δεν, το, δεν ήθελε να το κάνει αυτό, την αμυψισφορά, αμυψισφορά συγγνώμη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή η ποικιλομορφία των καλλιεργιών ε, εφαρμόζεται σωστά ε, να μην πρέπει τελικά να καλλιεργούν ένα προϊόν οι ε, γεωργοί χωρίς τελικά να ανταμείβονται γι' αυτό γιατί βασίζονται σε κάποιο κανόνα θα αλλάξει αυτό, θα προσαρμοστεί δεόντως. Ε, τώρα για την τροφιμική αλυσίδα θα κάνετε, θα έχετε κάποια πρωτοβουλία ξεχωριστή για το θέμα του εφοδιασμού σε τρόφιμα, της αλυσίδας εφοδιασμού σε τρόφιμα ή θα συμπεριληφθεί σαν ένα κομμάτι τη κοινή αγροτικής πολιτική θα μετατραπεί, θα αλλάξει. Σας ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι για τις ερωτήσεις σας. Ολοκληρώσαμε τον κατάλογο των ομιλητών και θα δώσω το λόγο πάλι στον Επίτροπο για τις απαντήσεις. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ελπίζω να μπορέσω να καλύψω όλες τις ερωτήσεις. Σητώ συγγνώμη τον προτέρων, να τα καταφέρω, θα κάνω ό,τι μπορώ. Κύριο Σάνι, έθεσα κάτι. Στο πρόγραμμα εργασιών εμφανίζεται ο εξυγχρονισμός και απλούστευση της ΚΑΠ και τονίζεται και η πρωτοβουλία για την αλυσίδα εφοδιασμού σε τρόφιμα. Όσον αφορά αυτή την πρωτοβουλία, απαντώ και σε άλλους που έθεσαν το θέμα, τώρα προσπαθούμε να συμμορφωθούμε με την καλύτερη νομοθεσία, τα διάφορα βήματα πρέπει να γίνουν έτσι έχουν τα πράγματα, αυτό που να κάνουμε τώρα. Συνεργαζόμαστε την κυρία Μπεκόφσκα και τους άλλους για αυτά τα θέματα. Σημειώνω λοιπόν ότι γίνονται τροπολογίες στο Omnibus. Ίσως να υπάρξουν κάποια προβλήματα που θα πρέπει να λυθούν στην κατάλληλη φάση. Εγώ δεν είμαι δεσμευμένο όσον αφορά τη διαδικασία. Πρέπει να ακολουθήσουμε από τη στιγμή που θα πετύχουμε αποτελέσματα που είναι επωφελή για το Γιώργο. Αν κάποιε αλλαγέ στο Omnibus γίνουν αποδεκτέ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ευπρόσδεκτε οι αλλαγέ. Έτσι μπορούμε να κινηθούμε. Εξίσου θα έχουμε ξεχωριστή πρωτοβουλία. Αντί για προτάσματα το 2020 για θεμητέ πρακτικέ για τα τρόφιμα. Τώρα, όσον αφορά για, τον, ε, για την πανόλη των χείρων, ο κ. Ανδρουκάητης εργάστηκε σκληρά, έδωσε και αρκετά χρήματα, δοθήκαν σε ανθρώπου, για να βοηθήσουμε την εκρίζωση τη ασθένεια και να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε του γεωργού να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα. Και οι χώρε που γνωρίζετε την περιοχή σα είναι στο επίκεντρο της προσοχής μας, κτηνοτρόφοι. Θέλουμε να εξαπλωθεί λιγότερο η ασθένεια, αλλά μόλι πρόσφατα το καταφέραμε αυτό. Το χείριο κρέα είναι πολύ σημαντικό για το εμπόριο σαν προϊόν. Και είχαμε μεγάλη επιτυχία στην Κίνα με αυτό το προϊόν. Με εξαγωγέ χειρίου κρέατος στην Κίνα. Δεν θέλουμε να έχουμε ασθένεια που δεν είναι, που θα είναι ανεξέλεγκτη και θα διασπαρεί σε άλλε χώρε όπω είναι η Ρουμανία, Πολωνία, Βουλγαρία και οι βαλτικέ χώρε. Παρακολουθούν προσεκτικότατα την κατάσταση για να προστατεύσουμε το εμπόριο. Όσον αφορά και άλλα χρήματα. Δεν έχουμε άλλα χρήματα δεν έχουμε, πρέπει να προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε του πόρου που έχουμε μέσω των μέτρων αναπτύξης υπαίθρου. Δώσαμε όλη την ευελιξία στα κράτη-μέλη να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν του πόρου, ούτω ώστε να μπορέσουν να αλλάξουν τα προγράμματα αναπτύξης υπαίθρου για να βοηθήσουν του γεωργού. Φλάνναγκαν, Ελπίζω να αντιμετωπίσω ε, με ρεαλισμό τα προβλήματα του Brexit και ο συναισθηματισμό. Και θα ξοδέψω πάνω από μισή ώρα. Εστέ βέβαιο. Φανταστείτε τι μου λένε πολλοί άνθρωποι έρχονται σε επαφή μαζί μου πάνω σε αυτό. Είναι πολύ δύσκολο και απογοητευτικό στα διαδικασία τώρα. Διότι δεν ξεκινήσαν καν οι διαπραγματεύσει. Δεν θα ξεκινήσουν μέχρι τα μέσα Ιουνίου. Αλλά όσο προχωρούν και ξέρουμε ποιο είναι το θεματολόγιο, η ατζέντα. Η ατζέντα είναι αρκετά καλή από πλευρά Δημοκρατία Ιρλανδίας. Αναγνωρίζεται από το Κοινοβούλιο και όλα τα θεσμικά όργανα ότι υπάρχει, υπάρχουν ιδιαίτερε περιστάσει που επικρατούν και αφορούν την Ιρλανδία και δεν ισχύουν αλλού, διότι έχουμε μια διαιρεμένη νήσο και έχουμε τι εμπορικέ σχέσει σχέσεις βορρά-νότου και ανατολή δυσης Αυτά είναι θέματα τα οποία αναγνωρίζονται από όλου και αυτό είναι πρόσδεκτο. Και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω πάντα έκανε, στήριξε την εθνική διαδικασία και την Συμφωνία Μεγάλη Παρασκευή, την υποστήριξε επί οικονομικό επίση και σίγουρα στις κατευθυντήριε γραμμές που δημοσιεύτηκαν από το Συμβούλιο στις 29 Απριλίου βλέπουμε ποια είναι η ατζέντα για το βραχυπρόθεσμο μέλλον. Έχουμε τα οικονομικά θέματα που θα επηρεάσουν το μέλλον ΚΚΑΠ, τα θέματα δικαιωμάτων πολιτών που αφορούν την ελευθερία της, ε, να ξέρουν πού βρίσκονται οι άνθρωποι στον διακίνησή τους, και μετά τα θέματα των συνόρων. Δεν αφορά την Ιρλανδία, αφορά την Κύπρο και την Ισπανία και το Γιβραλτάρ. Αυτά είναι θέματα προ επίλυση. Σα λέω λοιπόν ότι δεν θα επαναπαυθούμε στι δάφνε μα. Αυτό που θα κάνουμε θα είναι να ακούμε παρατηρήσει και σχόλια για την ώρα. Δεν είμαστε καν στην αφετηρία δυστυχώ. Σίγουρα με τα χαρά να σας ενημερώνω βάσει των εξελίξεων. Κύριε Ντεκάστρο, το Συμβούλιο πρέπει να λάβει θέση όσον αφορά το Omnibus δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα όσον αφορά τι απόψει του Συμβουλίου, τι θα κάνει το Συμβούλιο. Ελπίζω η Μαλτέζικη Προεδρία να μπορέσει να πετύχει κάποιο αποτέλεσμα στην κοίτα το μέλλον όσον αφορά το Συμβούλιο και τη θέση του. Είσαστε προπορεύεστε όσον αφορά αυτά που υποσχεθήκατε ότι θα κάνατε και αυτά που πετύχατε εσεί και ο κύριο Ντε στο Κοινοβούλιο. Και εμεί είμαστε έτοιμοι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κινηθούμε. Αναφέρθηκε άλλο για το θέμα των επικεφαλή εταιριών στην ανάπτυξη υπαίθρου, των μεγάλων εταιριών και πρέπει να στηρίξουμε τα προγράμματα ανάπτυξη υπαίθρου για να συμβούν πολλά περισσότερα και ταχύτερα και με μεγαλύτερη ευθύνη και υπευθυνότητα. Θα το κάνουμε αυτό και θα κάνουμε σχετικέ προτάσει και θα δούμε πώ μπορούμε να προσθέσουμε τα θέματα που αφορούν ε, ε, του κρατικού ε, διαγωνισμού για την ανάπτυξη τη υπαίθρου, για τα προγράμματα τη ανάπτυξη υπαίθρου και τα βιοκαύσιμα. Το ρώτησαν αυτό διάφοροι. Θα απαντήσω με τη μια. Επίτροπο Κανιέτα έκανε κάποιε προτάσει στα πλαίσια τη Ενεργειακή Ένωση και τα βιοκαύσιμα και οι στόχοι του 2020 αρχικά ήταν 7% για πρώτη γενιά, καύσιμα πρώτη γενιά. Το αποτέλεσμα ήταν 4,1% Χρήση ε, βιοκαυσίμων πρώτη γενιά. Και υπάρχει μια κίνηση για το 2030 προς προωθημένα βιοκαύσιμα και το στοιχείο που έχει προταθεί και προβληθεί για τους σκοπούς συζητήσεως από τους νομοθέτες είναι 3,8%. Οπότε έχουμε τη χρήση 4,1%, έχουμε προτάσει 3,8%, δεν απέχουμε πολύ, 7% ποτέ δεν επιτεύχθη και ποτέ δεν θα επιτευχθεί. Διότι η τεχνολογία κινείται γρήγορα προ τα προχωρημένα βιοκάψιμα. αλλά δεν μπορούμε να καταλήξουμε τα βιοκάψιμα τη πρώτη γενιά λόγω των επενδύσεων που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Και γι' αυτό θα ήταν πολύ άδικο για εκείνου από πλευρά πολιτική να το κάνουμε αυτό να αρχικά να κινηθούμε για βιοκαύσιμο από τι γενιέ και μετά να στραβήξουμε το χαλί κατά τα πόδια. Θα πρέπει σταδιακά να γίνουν οι αλλαγέ και ο Επίτροπο Κανιέται το εξετάζει αυτό στα πλαίσια των στόχων του 2030. Πρέπει να πω προ τον κύριο Νίκολα Καπούτα, το φίλο μου, ότι τα θέματα που θέσατε για την ξυλέλα αφορούν τον κύριο Ανδροκάητη. Αλλά θα με ενημερώσει πλήρω και θα σε ενημερώσω και εγώ με τη σειρά μου. Θα μιλήσω αύριο μαζί του για αυτό το θέμα. Δεν ξέρω ποια είναι η κατάσταση παρούσα όσον αφορά τα λεόδεντρα. Ξέρω ότι είναι πολύ ευαίσθητο θέμα για την Ιταλία, την περιοχή τη Πούλια και την Νότια Ιταλία εν γέννη. Από ό,τι καταλαβαίνω, κινείται λίγο προ βορρά πρόσφατα. Τέλο πάντων. Έχουμε ανησυχητικέ εξελίξει, άρα πριν καταλήξω κάποια συμπεράσματα για κάτι για το, το οποίο δεν γνωρίζω πλήρω, θα θέλω να συζητήσω με τον κύριο Ντρουκάητη για να ενημερωθώ πλήρω. Αύριο θα μιλήσω μαζί του. Η κυρία Τανσίλα, ε, έχουμε ίδια μέτρα στο σύστημα αυτό, στην παρούσα ΚΑΠ για την υποστήριξη μικρών εκμεταλλεύσεων. Είναι το πακέτο για τι μικρέ Δεν το χρησιμοποιούν όλε οι χώρε, ούτε κάθε περιφέρεια ή κάθε περιοχή. Και γι' αυτό εγώ θα υποστήριζα ένθερμα μια κλίση της υποστηρίξεως περισσότερο προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μικρομεσαίες εκμεταλλεύσεις, να επικεντρωθούμε από αυτόν, αν έχουμε προβλήματα για τον επόμενο γύρο των καταρτήσεων του προπολογισμού. Τα κονδύλια θα κάνουν τη διαφορά. Σε αυτό, αλλά σίγουρα το θεωρώ το θέμα της μελλοντική χρηματοδοτήσεως. Δεν το υποστηρίζω αυτό. Όσον αφορά τη σύγκληση, αυτά είναι θέματα που αφορούν το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Δεν μπορώ να απαντήσω σε ερωτήσει τώρα. Δεν έχω ιδέα ποιο θα είναι ο προπολογισμό. Δεν ξέρω περισσότερο από εσά ούτε κανένα άλλο. Από τη στιγμή που θα έχουμε σαφήνει σε αυτόν τον προπολογισμό, θα μπορέσουμε, ελπίζω, να πολεμήσουμε, να δώσουμε τη μάχη μα για ισχυρή ΚΑΠ που θα είναι καλά χρηματοδοτημένη. Τώρα τα βιολογικά προϊόντα. Έχουμε 95% του θέματο και θα ενημερωθείτε. Έχουμε 4-5 μεγάλα προβλήματα προ επίλυση, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αναφέρθηκαν από του φίλου μα από τη Φιλανδία και τη Σουηδία. Ξέρω ότι είχατε πολλέ συναντήσει σήμερα. Δεν περιμένετε μέσω ανακοινωθέντων τύπου τύπο να διαπραγματευτώ. Δεν θα το περιμένετε κάτι τέτοιο. Δεν θα αντιδρούσατε σε ανακοινωθέν τύπο. Αλλά μπορώ να σα πω ότι είμαστε πολύ ευαίσθητοι όσον αφορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε και που αναφέρατε όσον αφορά τα θερμοκήπια. Και τα θέματα είναι πάρα πολύ είναι πασίγνωστα. Τα ξέρει ο κ. Χάουζινγκ. Οπότε ελπίζω να μπορούμε να συνεργαστούμε, ώστε να καταλήξουμε σε μια λογική λύση, ώστε να λάβουμε υπόψη τι ιδιαίτερε ευαισθησίε. Είναι ένα ευαίσθητο θέμα, ευαίσθητο τομέα και το δεχόμαστε αυτό, το παραδεχόμαστε χωρί κάποια επιφύλαξη α, του τελικού αποτελέσματο. 31 Μαου είναι άλλωστε με διαλόγο. Κύριε Χάουφμαν, είσαστε εντάξει 7 Μαου. Το Ευρωκοινοβούλιο δεν, δεν συνεδριάζει. Είναι Παρασκευή και από ό,τι λέει ο Πρόεδρο θα μπορέσετε να παραστείτε στι Βρυξέλλε. Είσαστε εντάξει. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη έχετε συνεδριάσεις. Ελπίζω ε, να δεχτείτε ότι το ελέγξαμε. Είναι θαύμα που έγινε, αλλά όπως είπε ο Πρόεδρος, είμαστε εντάξει πάνω σε αυτό. Υπάρχουν πρακτικά ζητήματα όμως που υπάρχουν και περιστρέφονται γύρω από τη στέγαση για 500 ανθρώπους και μετάφραση. Ε, ξέρετε, δεν θα καταφέρουμε να ικανοποιήσουμε όλου όσον αφορά το πού θα στεγαστούν. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να του ικανοποιήσουμε όμω. Και μα λέει ο Πρόεδρο ότι τα πάντα είναι εντάξει. Και σίγουρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτή η Επιτροπή θα εκπροσωπείται και θα στηρίξει τι θέσει τη. Άριστα. Δεν κατάλαβα την ερώτηση που θέλατε να θέσετε. Ίσως να το κουβεντιάσουμε μετά. Δεν έπιασα το ερώτημά σας. Δεν θα απαντήσω μια ερώτηση που δεν ερωτήθηκε. Μήπω διμερώ, αν μπορούμε να το λύσουμε, μετά να συναντηθούμε για να πιάσω καλύτερα την ερώτηση που θέσατε. Ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν κατάλαβα. Για του ενεργού καλλιεργητέ του Omnibus δίνουμε δυνατότητα στην πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχουμε περιοχέ και κράτη-μέλη που θα αποφασίσουν από αυτού όσον αφορά τον ορισμό του ενεργού καλλιεργητού. Δεν πετύχαμε ομοφωνία ή καλό αποτέλεσμα. Α, όλοι αισθάνθηκαν κάπως ε, ανικανοποιητοί την περισμένη φορά. Είχαμε αρνητικό κατάλογο, αντίθετικό κατάλογο, να δούμε τι πρέπει να κάνει και τι θέλει να κάνει η κάθε χώρα και κάθε περιοχή στα πλαίσια της επικουρικότητας. Τι θέλει να κάνει κανείς, γιατί είναι επίμαχο θέμα. Για το αντιντόμπινγκ, για τις πατάτες από τη Βραζιλία δεν το ήξερα. Ίσως να είναι ο ειδικό σας τομέας στο Βέλγιο, ίσως μπορείτε να με ενημερώσετε. Γι' αυτό δεν το ήξερα με τα χαράς να ακούσουμε αν υπάρχει πρόβλημα. Ίσως να σας δώσουμε και κάποιες, να μου δώσετε λεπτομέρειες για τους νέους καλλιεργητές. Σε όλες τις παρεμβάσεις εδώ και αλλού ανέφερα την ανανέωση των γενναιών. Είναι κάτι που πρέπει να επεξεργαστούμε, να εργαστούμε σκληρά. Να θέλουν οι νέοι να παραμείνουν στη Γεωργία όχι μόνο αυτοί που ανακατεύονται με τι καλλιέργειε, αλλά στι άλλε επιχειρήσει σχετιζόμενε με τη γεωργία και να δημιουργηθούν θέσει εργασία στην Ήπεθρο μέσω έρευνα, καινοτομία, περαιτέρω υποστήριξη, ήπια νομοθεσία, χρηματοπιστωτικών μέσων, να βοηθήσουμε του νέου να παράξουν νέε επιχειρησιακέ ευκαιρίε στον τομέα τη γεωργία. Με τα χαρά το κάνουμε αυτό, όπω ανέφερα, και τι πρακτικέ αθέμητε εμπορικέ πρακτικέ το ανέφερα και αυτό. Θα μάθουμε από την εμπειρία τη Κροατία. Τι κάνετε για του νέου ε, γεωργού. Κυρία Ελπίζω ότι έχετε καλά γυαλιά. Μην με πυροβολείτε όμως. Συμφωνώ. Μην με πυροβολήσετε, αλλά συμφωνώ με αυτά που είπατε. Γι' αυτό εξυγχρονούμε την ΚΑΠ, εξυγχρονίζουμε την ΚΑΠ. Διότι μετά την τελευταία μεταρρύθμιση του 2013 είχαμε συμφωνία των Παρισίων, έχουμε στόχου βιώσιμη αναπτύξεω, συμπεφωνημένου στόχου και δεν θα πρέπει να έχουμε τι συμφωνίε, να τι συνάπτουμε και να μην κάνουμε τίποτα. Επίση, κάναμε σημαντική πρόοδο, και εδώ παντούμε στην ερώτηση τη κυρία Ρόκερ. Κάναμε σημαντική πρόοδο σχετικά με τα εμπορικά ζητήματα δεν υπάρχει αντιντόμπινγκ για τα εμπορικά. Δεν υπάρχει ντόμπινγκ γεωργικών προϊόντων στην Αφρική. Αυτό είναι κάτι που απασχολεί ιδιαίτερα τα ΜΜΕ. Καμιά φορά σε γερμανικά τηλεοπτικά προγράμματα δεν βλέπουμε αυτά. Και εκεί του παρουσιάζω ποια είναι η πραγματική θέση. Και δεν θέλουν όμω να διαβιβάσουν τη θέση, τη σωστή, την πραγματικότητα, όπω να ανακοινώνω εγώ. Παίρνουμε χωρί δασμού διάφορα προϊόντα από χώρε ΑΚΕ, από την Αφρική, αδεσμολόγητα. Είμαστε η μόνη περιοχή, η χώρα που έχει γίνει αυτό και έχουμε τον Αιρόμπι συμφωνία για, τον, για την κατάργηση ε, επιδοτήσεων σε εξαγωγέ, κάτι που ισχύει για όλε τι ευρωπαϊκέ χώρε. Από 1η Πρώτου 2016 ηγήθηκε η Ευρώπη στον αφορά το θέμα αυτό. Νομίζω ότι έχουμε πολλά θετικά στοιχεία για τα θέματα αυτά που αναφέρατε και ελπίζουμε στο τέλο τη διαδικασία για τον εξυγχρονισμό τη ΚΑΠ θα δούμε περισσότερα θετικά αποτελέσματα. Ξέρουμε, ξέρουμε. Έχουμε πείχνει του γεγονότο. Είναι απαράδεκτο να καταστρέφουμε τις τοπικές αρχηγές στο Μαλί ή σε οποιαδήποτε άλλη αφρικανική χώρα. Καμιά φορά καθορίζουν τις τιμές τους για δικούς τους εσωτερικούς σκοπούς, για τους ντόπιου παραγωγούς, του, ώστε να μπορούν να επιβιώσουν. Η Ευρώπη όμως δεν κάνει κάποια συνεισφορά στον αφορά αυτό το ντάμπινγκ. Ίσως να το έκανε κατά το παρελθόν, αλλά δεν το κάνουμε τώρα. Τώρα, στον αφορά είπε η κυρία Μαγκίνες θέλω να γίνει ποια αξιολόγηση του, της υπόψη του πρασινίσματος της Γεωργίας, να λάβουμε υπόψη τα θέματα του περιβάλλοντος και στι δίποτε πρωτοβουλίε που θα διαφανούν θα προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα τη ποικιλομορφία των καλλιεργιών. Ε, το θέμα επίση τη απόδοση των καλλιεργιών, ε, μόνιμων βοσκοτοπιών, βοσκοτοπίων κλπ. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το αναλύσουμε. Είναι πολύ δύσκολο, εξαρτάται από τα κράτη-μέλη. Αν θέλουμε να πετύχουμε του στόχου στην αλλαγή του κλίματο και του στόχου που έχουμε θέσει και τη συνεισφορά που μπορεί να κάνει η Γεωργία σε αυτού του σκοπού, ίσω πρέπει να λάβουμε δύσκολε αποφάσει. Αλλά τουλάχιστον προσπαθήσουμε να δούμε το πρασίνισμα τι έχει πετύχει μέχρι τώρα. Και θα κάνουμε την αξιολόγηση μέχρι το τέλο του έτου. Και ελπίζω ότι θα διεξαχθεί μια καλή συζήτηση από αυτού που προανέφερα ότι έχουμε ξεχωριστό θέμα τη αλυσίδα των τροφίμων και κάποια θέματα για το όμνιμπους. Κυρία Ριμπέρο, σίγουρα θα προτιμούσαμε να μην ξανανοίξουμε ε, το άλλο θέμα το πρόγραμμα ΠΟΖΕΙ δεν θέλουμε να το ξανανοίξουμε. Ήδη όμως κάνουμε τις σωστές προσαρμογές για τις περιοχές ΠΟΖΕΙ για να έχουμε συμπληρωματική στήριξη πέραν ε, των πόρων για την άξιση πέθρου. Εκτός μικροφώνου, έξω το μικρόφωνο του κύριου Πιτρόπου, τον ακούμε. Μερικές φορές οι περιφέρειες ε, δεν αξιοποιούν την ελαστικότητα που έχουν. Αλλά όποια περιφέρεια, ακόμη και οι Αζόρες, ε, επιθυμούν να αλλάξουν το πρόγραμμα από μπορούν να το κάνουμε σε δύο μήνε, αν θέλουν να δώσουν περισσότερη έφαση σε μία περιφέρεια ένα τη άλλη. Υπάρχει δυνατότητα, υπάρχει τέτοια ελαστικότητα για σημαντικέ αλλαγέ. Νομίζω ότι υπάρχει αρκετή ευελιξία στο ΠΟΣΕΙ. Μπορεί να διαφωνείτε, αλλά κατά τη γνώμη μου είναι αρκετή ελαστικότητα που εξασφαλίζει το πρόγραμμα ΠΟΣΕΙ. Ο κύριο Γιάννη είπε ότι μόνο πέντε χώρε ε, έχουν δώσει απαντήσει για την ΚΑΠ. Όχι, δεν σα έχουν ενημερώσει σωστά. Και 28 χώρες μέλη έχουν στείλει απαντήσεις, αλλά η Γερμανία πραγματικά έχει, έδωσε πολλές απαντήσεις. Κάποιος ε, ενεργοποιήθηκε στη Γερμανία και στους επίπεδο παραγών και με κυβερνητικών οργανώσεων και ήταν ε, πάρα πολλά τα σχόλια από τη Γερμανία. Πάντως ε, οι περισσότερες απαντήσεις όντως δόθηκαν από τη Γερμανία αλλά όλες οι χώρες έστειλαν απαντήσεις. Η παραγωγή πρωτεΐνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ανέκαθεν ελληματική και δεν υπάρχει καμία ελπίδα να καλύψουμε αυτό το κενό, γιατί δεν είμαστε ανταγωνιστικοί ούτε με τις ΗΠΑ ούτε με τη Λατινική Αμερική. Υπήρχε μια μικρή αύξηση των πρωτενούχων καλλιεργιών τα τελευταία χρόνια, αλλά υπήρχε ακόμη μεγαλύτερη αύξηση των ε, εισαγωγών. Και φυσικά υπάρχουν εθελοντικές συνδεδεμένες ενισχύσεις ε, και στη Γερμανία μπορείτε να τις αξιοποιήσετε για να προωθήσετε τις πρωτεϊνούχες παραγωγές, μακάρι εκτός των χώρων οικολογικής εστίασης, θα το προτιμούσα. αλλά το θέλετε εντός των χώρων ε, οικολογικής εστίασης, χρειάζεται και πλέον μέτρα για να προστατεύσετε τη βιοπικιλότητα που επίσης είναι πολύ σημαντική. Και 30% του προϋπολογισμού πηγαίνει στο, στην ε, οικολογικοποίηση της γεωργίας, στο πρασίνισμα που λέμε, γιατί θα πρέπει να τηρήσουμε τις υποσχέσεις που δώσαμε για το 2030 και συμβάλλουμε και εμείς αυτή την τηρήση των στόχων. Φυσικά η απλούστευση είναι προτεραιότητα και όντω έχουν εκνευριστεί πολλοί γεωργοί με το επίπεδο πολυπλοκότητας της εφαρμογής της ΚΑΠ και αυτό το πρόβλημα θέλουμε να το διορθώσουμε. Βέβαια δεν πρόκειται να γίνει εν μία νυχτή γιατί θα πρέπει να αλλάξουν κάποιες, κάποιοι βασικοί κανονισμοί. Ε, πάντως ε, έχουμε μια δέσμη μέτρων ε, για τους ελέγχου τον Ιούλιο για να δείξουμε πώς οι νέε τεχνολογίες μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο αντί να έχουμε ε, τις επιτόπιους ελέγχους και να χάνουν έτσι πάλι το χρόνο τους ε, όταν μπορούν να, να υιοθετήσουν άλλες μεθόδους και να μην δημιουργήσουμε αυτό το, κλίμα φόβου. Επίσης έχουμε ε, προληπτικούς ε, ελέγχους, προκατακτικούς, ώστε να μπορεί ο υπάλληλος να ελέγχει εκ των προτέρων το, την αίτηση να δει σωστή και αν υπάρχουν μικρολάθη να διορθώνονται εγκαίρως, ώστε να μπορεί ο Γεωργός να υποβάλει τελική του έκθεση, ε, την τελική του αίτηση χωρίς να έχει λάθη που θα καθυστερήσουν ώστε να μην έχουν την πίεση οι Γεωργοί και να ξέρουν ότι από τη στιγμή που η αίτησή του είναι σωστή, κατά πάσα πιθανότητα θα λάβουν και τα κονδύλια. Όντω, πολλοί Γεωργοί βρίσκονται στη Ρουμανία και είναι η Ρουμανία έχει γεωργικό κλάδο εντάσσεω εργασίας, αλλά πιστεύω ότι θα κάνουμε κάποιες απλουστεύσει για να κάνουμε ευκολότερη την πρόσβαση των γεωργών. Και για, για τα πουλερικά ελευθερία βοσκή θα υποβάλουμε κάποιες προτάσεις, θα ελέγξω ε, τι νομικές προτάσεις και θα επανέλθω για να σας δώσω πιο ακριβείς απαντήσεις. Η κυρία Ρασκαρσία εντυπωσιάστηκε από το χρονοδιάγραμμα του εξυγχρονισμού της ΚΑΠ. Θα πρέπει να συνεχίσουμε πάντως το έργο μας, παρόλο που ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα προϋπολογισμού που δεν πρόκειται να επιληθούν και ίσως και μάλλον θα υποβάλουμε την ανακοίνωση υπό την επιφύλαξη της μελλοντική διαμόρφωσης του προϋπολογισμού. Και ελπίζω να βληθούν ε, τελικά τα προβλήματα, παρόλο που δημοσιονομικά προβλήματα δεν θα θα συνεχίζουν να μας ταλανίζουν για μια διετία ακόμη. Μίλησα για τις νέες αγορές, τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Έχουμε το θέμα της ασφάλειας των τροφίμων, της αύξησης του πληθυσμού, του εμπορίου και πώς θα εξασφαλίσουμε και μια βιώσιμη παραγωγή. Γι' αυτό και θέλουμε εξυγχρονισμό της γεωργίας, περισσότερες δράσεις για το περιβάλλον, εξασφάλιση της βιωσιμότητας. Δεν θέλουμε να παρακάμψουμε αυτούς τους στόχους. Και εναπόκειται και στους νομοθέτες ε, να προσαρμόσουν τις προτάσεις μας ώστε να λαμβάνουν υπόψη και τους στόχους αυτούς. Με εξαίρεση την ερώτηση της κυρίας Χούιμποχ που δεν την κατάλαβα καλά, νομίζω ότι τις υπόλοιπες απάντησα κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν κάποιος ε, συνάδελφος ε, δεν θεωρεί ότι απαντήθηκε πλήρως η ερώτησή του και έμεινε κάποιο κενό να ζητήσουμε ενδεχομένω γραπτή συμπλήρωση των απαντήσεων. Άλλωστε αυτό το συνηθίζουμε, είναι πια πρακτική της Επιτροπής. Σε ό,τι αφορά τις διαβουλεύσεις, οι διαβουλεύσεις δεν ολοκληρώθηκαν. Ε, οι διαβουλεύσεις ε, έχουν μια συνέχεια. Βέβαια μπορεί να ολοκληρώθηκε ένα στάδιο και να περάσουμε στο επόμενο στάδιο, αλλά οι διαβουλεύσεις ε, είναι μια αέναη κατάσταση. Επίσης έχουμε κάποια ε, σοβαρά προβλήματα τώρα και έχουμε και πρόβλημα πώς θα διαμορφωθεί μελλοντικά η κοινή πολιτική. Γιατί ταυτόχρονα προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τις τρέχουσες κρίσεις και να διαμορφώσουμε τη μελλοντική κοινή, πολιτική. Ε, θα έχουμε στο μεταξύ και τον Brexit, επιπλέον δυσκολία. Σου και πολλές ερωτήσεις περιστράφηκα γύρω από αυτό το θέμα. Επίσης, γνωρίζουμε από τους δικούς μας γεωργούς ότι ε, περιμένουν πολλές λύσεις από τους πολιτικούς γιατί ξέρουν ότι οι πολιτικοί επηρεάζουν την κατάσταση και ε, η πολιτική φυσικά επηρεάζει και την κοινή γεωργική πολιτική. Αυτά σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την ανταλλαγή απόψεων. Ολοκληρώνουμε το διαρθρωμένο διάλογο και περνάμε στο επόμενο σημείο. Ε, ελπίζω να μην προσβληθεί ε, ο, δε, μάλλον, κύριε Επίτροπε, δεν προσβληθούμε αν παραμείνετε στη συζήτηση και ακούσετε την ενημέρωση από τον κύριο Χόισλικ. Το αντίθετο, θα μείνουμε και ικανοποιημένοι αν παραμείνετε στην συνεδρίασή μας. <clears throat> Κύριε Πρόεδρε, δυστυχώς ο Επίτροπος δεν έχει χρόνο, αλλά θα είμαι σύντομος εγώ. Στον τελευταίο τριμερή διάλογο, το 17ο, είσαστε από την αρχή παρόν και τονίσατε την σημασία ε, ε, που αποδίδουμε στον προηγούμενο τριμερή διάλογο και είδατε και ο ίδιος κύριε Πρόεδρε πόσο δύσκολα ήταν τα θέματα των λεπτομεριών και η επίτευξη συμβιβαστικών λύσεων και πόσο δύσκολα είναι ακόμα τα πράγματα. Έχουμε ένα τριμερή διάλογο μπροστά μας και είμαστε αποφασισμένοι αν, όταν από την πλευρά μας, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρήσουμε ότι οι θέσεις μας καλύπτονται να ολοκληρώσουμε αλλά ε, πολλά μέλη να γίνουν μέχρι εκεί αν, θα αναφερθώ στα τέσσερα σημεία που συζητούνται ακόμη ε, πρώτον ότι ως Κοινοβούλιο εμείς θέλουμε μια ρύθμιση για τους σπόρους στα βιολογικά Θέλουμε ε, να τακτοποιηθεί η αγορά και να ρυθμίσουμε ε, το ε, υλικό των σπόρων που είναι πολύ ετερογενές. Επίσης από το Συμβούλιο δεν προβλέπονται εξαιρέσει για το βιολογικό τομέα. Ε, βέβαια έχουμε δεχτεί ότι θα λήξουν οι εξαιρέσει κάποια στιγμή και ε, οι σπόροι πρέπει να ε, φτάνουν στην αγορά. Εμείς ως Κοινοβούλιο υποβάλαμε την τελευταία φορά μια πρόταση και πιστεύω ότι αν υπάρχει καλή θέληση θα καταλήξουμε σε αποτέλεσμα. Πάντως είναι πολύ σημαντικό να, για το Κοινοβούλιο να βρεθεί η ρύθμιση εδώ. Για τις βάσεις δεδομένων έχουμε συμφωνήσει σε μεγάλο βαθμό. Για τους σπόρους ε, θέλουμε να δημιουργήσουμε βάση δεδομένων για όλα τα κράτη-μέλη ούτως ώστε όλοι, όλες οι ομάδες ε, παραγωγών να ξέρουν για τους σπόρους. Εκεί που δεν συμφωνούμε είναι πότε η ε, ε, άδειες ε, που προβλέπουν εξαιρέσεις θα λήξουν. Είχε πει αρχικά η Κομισιόν το 2021, πράγμα που δεν θεωρείται ρεαλιστικό. Τώρα συζητάμε για 15 χρόνια μετά την έναρξη σε, με τη θέση σε εφαρμογή του κανονισμού. Ε, για τον οικολογικό τομέα υπάρχει και ε, η εθελοντική βάση. Ε, χρειάζεται αυτό, πρέπει να υπάρχει μια ευελιξία. μπορεί να συμφωνήσει το Κοινοβούλιο εδώ. Επίσης η στρεματική ενίσχυση και τα θερμοκήπια ήταν άλλο θέμα. Διευκρινίζω για εκείνους που δεν το γνωρίζουν ότι δόθηκε μεγάλη μάχη γιατί υπήρχε το σχέδιο ε, της Κομισιόν που δεν προέβλεπε εξαιρέσεις. Ε, υπάρχει μια εξαίρεση στον τωρινό κανονισμό για 20-30 ε, εκτάρια ε, στις σκανδιναβικές περιοχές στη Βόρεια Ευρώπη από την έκθεση Hector ε, που αξιολογήθηκε και τώρα πολλές καμιναδικές, ε, πέντε ε, χώρες βόρειες είπαν ότι για λόγους κλιματικούς θα πρέπει να, η παραγωγή αυτή να επεκταθεί προς νότον. Αυτό μπορεί να γίνει, αλλά όταν διαπιστώσουμε ότι στο, στα πλαίσια της Ένωσης ε, δεν θα έχουμε μια παραγωγή όπου δεν θα είναι ο κανόνας η θεματική παραγωγή. μεταξύ Νότιας Δανίας και Βόρειας Γερμανίας δεν υπάρχει κλιματικό όριο. Οπότε είναι δύσκολος ο διαχωρισμός και όταν μιλάμε για στρέβλωση του ανταγωνισμού ε, είναι δύσκολο να πούμε ότι υπάρχει στραματική ε, παραγωγή στη Δανία ενώ στη Γερμανία δεν υπάρχει. Υπάρχει δηλαδή φόβος ότι μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα. Ή θα ε, περιοριστούμε στον 62ο παράλληλο ή θα χαράξουμε ένα μεγαλύτερο κύκλο για να καλύψουμε τις 5-6 χώρες που έχουν πρόβλημα ε, Φιλανδία, Σουηδία, Δανία, οι σκανδιναβικές χώρες αλλά εκεί θα ε, υπάρχουν μεγάλες ε, μειώσεις στην παραγωγή. 80% είναι η δική μας πρόταση ούτως ώστε να παραμείνει εξαίρεση το σύστημα αυτό. Ένα άλλο θέμα είναι οι οριακές τιμές στα παρασιτοκτόνα. Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο συμφωνούν εδώ ότι οι οριακές τιμές δεν, που προτείνει η Κομισιόν δεν γίνονται αποδεκτές. Υπάρχουν όμως τρεις χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν αυτές τις οριακές τιμές Οπότε μάλλον θα υπάρξει συμβιβαστική λύση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταρχήν δεν θα αλλάξουμε τίποτα έως ότου υποβάλει την έκθεσή της η Κομισιόν για την κατάσταση αυτή, δηλαδή από πού προέρχονται οι ρήποι, ε, τι εύρος έχουν και πώς αντιμετωπίζονται. Θα δούμε αν το 2022 θα τα ξαναδούμε όπως θέλει το Κοινοβούλιο ή το 25 όπως θέλει το Συμβούλιο αν θα ε, πρέπει να ε, αναθεωρηθεί αυτή η έκθεση της Κομισιόν. Δεν θέλουμε δηλαδή τροποποίηση του καθεστώτος μέχρι τότε. Το αν θα τα καταφέρουμε θα το δείξουν οι μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Αυτά είναι τα τέσσερα σημεία τα οποία συζητούνται ε, θα πρέπει να βρεθούν λύσεις ε, ανάμεσα στα ε, τρία θεσμικά όργανα και εμείς πρέπει να κάνουμε συμβιβασμούς αλλά νομίζω ότι βρέθηκε μια βάση. Ο Επίτροπος είπε 95% έχουν συμφωνηθεί τα θέματα, κατά 95% είπε, νομίζω κατά 90% έχουμε τελειώσει. Υπάρχουν και ορισμένα άλλα θέματα ε, ένα άλλο που εμάς μας φαίνεται πολύ σημαντικό ε, δηλαδή οι ε, εταιρείε που παρασκευάζουν βρεφικές τροφές η πρόταση είναι να είναι πολύ αυστηρή η νομοθεσία αλλά ε, δεν θα μπορούσε να υπάρχει βιολογική παραγωγή ε, βρεφικών τροφών ε, έτσι. Οπότε αυτό δεν το δεχόμαστε. Θα πρέπει να δούμε τι συνέχεια θα δοθεί για να μην περιοριστεί αλλά να αναπτυχθεί στο μέλλον ο κλάδος. Αυτά είναι τα θέματα τα σημαντικά που πρέπει να τα λύσουμε μέσα από ένα συμβιβασμό. Ε, εν προκειμένου το Συμβούλιο είναι στο πλευρό μας, θα βρεθεί πρακτική λύση. Υπάρχουν και άλλα ανοιχτά θέματα τα οποία θα τα ε, συζητήσουμε στον τελευταίο τριμερή διάλογο αλλά είναι εφικτό να βρεθεί μια λύση και να φτάσουμε σε συμφωνία. Θα το κρίνουν ε, οι συνάδελφοι αν η καλή δουλειά που κάναμε ε, αρκεί για μια συμβιβαστική λύση ή όχι. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ε, έχετε πραγματικά πολύ δύσκολο έργο. Γιατί ε, η Προεδρία σηκώνει τα χέρια, χαμογελάει ευγενικά και λέει δεν έχουμε εντολή για αυτό το θέμα. Οπότε βλέπουμε ότι η Μαλτέζικη Προεδρία δεν είναι σε θέση να κάνει παραχωρήσεις που αυτό θα περιμέναμε και αυτό ελπίζαμε. Παρ' όλα αυτά, εγώ κρατάω την αισιοδοξία μου και ελπίζω στις 22 Μαΐου, σε μια εβδομάδα που θα γίνει ο επόμενος διάλογος, να έχουμε κάποια πρόοδο. Αλλά η εντολή είναι έτσι διαμορφωμένη που έχει δέσει τα χέρια της Προεδρίας, η οποία δεν έχει καμία ευελιξία και ελαστικότητα στο διάλογο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Ο Μάρτιν Χόισλιγκερ παρουσίασε τα επιμέρους θέματα ήδη. Πιστεύω ότι ο Επίτροπος ε, προηγουμένως ε, ξέφρασε υπερβολική αισιοδοξία ε, ότι 55% τα θέματα μάλλον 89 και 90, ε, έως 90% έχουν λυθεί. Άρα έχουμε δουλειά ακόμα μπροστά μας. Πολλά έχουμε καταφέρει. Και ο πρόεδρος ε, με πρόλαβε ήδη όταν είπε ότι είναι δύσκολο ε, μετά από μια αδιέξοδη κατάσταση όπως πέρσι με την προηγούμενη προεδρία να περάσουμε 3,5 μήνες για να μιλάμε για τα διαδικαστικά με την Προεδρία η οποία έρχεται με μια εντολή αυτό έγινε το, το Φεβρουάριο και τότε παρουσίασε την εντολή ως ε, μη ε, τροποποιήσιμη εγώ ε, άλλα πράγματα είχα μάθει ότι στις διαπραγματεύσεις ο ένας προσεγγίζει τον άλλον και δεν παρουσιάζει θέσεις που δεν επιδέχονται τροποποιήσεων. Πάντως χρειάστηκε αν κάποιες βδομάδες για να υπάρξει κάποια μετακίνηση. Και είναι θεμητές οι ερωτήσεις των ε, συναδέλφων ότι τι κάνετε εσείς εκεί στις διαπραγματεύσεις. Πάντως το τελευταίο διάστημα έγινε πρόοδος και είναι πάρα πολύ πιθανό ε, στον τελευταίο τριμερή διάλογο στις 31 Πέμπτου να ε, βρούμε λύσεις και να δούμε ότι και η Κομισιόν σε ορισμένα θέματα δεν ε, εξακολουθεί να έχει τόσο σκληρή θέση για τα φυτοφάρμακα κλπ. Μπορούμε λοιπόν με κάποιο με κάποια ε, αισιοδοξία ε, να ε, προχωρήσουμε προς τον τελευταίο τριμερή διάλογο ελπίζοντας ότι θα υπάρξει αποτέλεσμα. Ευχαριστώ κύριε Σαντρία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον Μάρτιν καταρχάς για τη δουλειά που έκανε σε αυτή την προσπάθεια που είναι περιπλοκότατη σαν θέμα. Στον τριμερή διάλογο είδατε πόσο περίπλοκα ήταν τα πράγματα για να προχωρήσουν διαπραγματεύσει. Το πρόβλημα στο τριμερή διαλόγου είναι ότι είμαστε τρει. Πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Μαρτίν Όσλινγκ γιατί από την αρχή τηρεί στεναρά και εφαρμόζει την εντολή του Κοινοβουλίου και σέβεται την ψήφο που έχει στην Επιτροπή βλέπουμε ότι η Προεδρία, ανάλογα με τις Προεδρίες, προχωρά σε κάποιες πτυχές σε σχέση με την προηγούμενη και κάνει επαναχωρήσεις. Και τώρα ξαναμπαίνουμε στην πρόοδο. Αλλά είναι κάπως αργά να προχωρήσουμε αυτό το θέμα. Αυτό που ισχύει για την Προεδρία ισχύει για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και λυπούμε που ο ο κύριος Χόγκαν δεν, δεν έμεινε, διότι όσον αφορά το θέμα των σπόρων έχουμε πολύ ακριβή προσέγγιση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της DG Sanko, συγγενικής θητής Sanko, να ανακρούει πρίμναν. Και πριν τον προτελευταίο τριμερή διάλογο είχαμε αντίθετη θέση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί το σημαντικού θέματος όπω είναι των σπόρων. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειε. Θα πρέπει να είμαστε αυστηροί στη θέση μα και αν μπορείτε να συμμετάσχετε στον επόμενο τριμερή διάλογο, να το πείτε όταν υπάρχουν θέσει που λαμβάνονται σε ένα χαρτοφυλάκιο, δύσκολα μπορούμε να πιστοχωρούμε και να επαναχωρούμε. Διότι αλλιώ υπάρχει κάποια βούληση να μην καταλήξει κάπου το θέμα αυτό για την προστασία των καλλιεργητών βιολογικών προϊόντων. Περιμένει ο τομέα διακαώ κάποιο αποτέλεσμα από τη συζήτηση και κυρίω όσον αφορά του πόρου. Πώ να το πω. Δεν θα πρέπει να επαναχωρήσουμε και θα πρέπει να παραμείνουμε στη θέση μα. Θα πρέπει τώρα να είναι διαθέσιμο ετερογενές υλικό για εκείνον που θα το χρησιμοποιήσει, κάτι το οποίο δεν ισχύει σήμερα. Πρέπει να διατηρήσουμε, διαφυλάξουμε τη θέση μας, διότι διαφυλάσσει τη βιοπικιλότητα, κάτι δεν είναι απλό. Παρόλο που έχω ελπίδε ότι θα καταλήξουμε κάπου, πρέπει να πω ότι το αριθμό των θεμάτων είναι τόσο μεγάλο. Πρέπει να ρυθμίσουμε τα περισσότερα θέματα πριν τον επόμενο τριμερή διάλογο. Διαφορετικά δεν θα καταλήξουμε τελικά στου σκοπού μα στον επόμενο τριμερή διάλογο. Ευχαριστώ κύριο Στάκουλα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ κύριε Χόισλινγκ, την ε, προηγούμενη εβδομάδα συναντήθηκα με Φιλανδούς παραγωγούς ε, βιολογικών προϊόντων θερμοκηπίου στις Βρυξέλλες. Μου είπαν ότι έχουν παγώσει όλες τι επενδύσεις ε, στον κλάδο αυτό και οι παραγωγοί αμφιβάλλουν ε, αν ε, θα επιβιώσουν ε, και θεωρούν ότι η Βρυξέλλες δεν θα πρέπει να περιορίζει τη βιολογική παραγωγή, αντίθετα να την προωθεί παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζω ότι στον επόμενο τριμερή διάλογο θα καταλήξετε σε μια ικανοποιητική λύση. Αντιλαμβάνομαι ότι προσπαθούμε να θεσπίσουμε κάποιες εξαιρέσεις για τις σκανδιναβικές χώρες στον κανονισμό, αλλά η απέτηση κατά τα 80% να είναι τοπική παραγωγή, επίσης είναι κάτι που περιορίζεται στο βορρά. Οι λύσεις μονοπωλίου δεν ε, ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες αυτών των χωρών. Αν θέλετε πραγματικά να ε, επιβιώσουν οι βιολογικοί παραγωγοί στην Ευρώπη, θα πρέπει να διευκολύνεται και τους σκανδιναβούς ε, βιολογικούς παραγωγούς ε, να συνεχίζουν τη δραστηριότητά τους και να μην τους εξωθήσετε σε διακοπή των δραστηριοτήτων τους. Στη Φιλανδία έχουμε γόνιμα εδάφη που χρησιμοποιούνται και σε βιολογικά θερμοκήπια και έχουμε τα καλύτερα δυνατά υποστρώματα αλλά οι απαιτήσει που προτείνει η Επιτροπή είναι υπερβολικές και σε ό,τι αφορά τις μικρές γλάστρες δεν υπάρχει κανένας περιορισμός σε ό,τι αφορά το, την ποιότητα του χώματος. Δεν είναι λογική η πρόταση. Όσο μεγαλύτερη είναι η γεωργική εκμετάλλευση, τώρα υπάρχει η, η απέτει το 80% του χώματος να προέρχεται από την περιοχή, ενώ για τις μικρές γλάστρες, ε, τα μικρά υποστρώματα δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Είναι άδικο αυτό. Προσοχή λοιπόν, δεν θα πρέπει να περιορίσουμε υπερβολικά α, ε, τους ε, βιολογικούς γεωργούς. Θα πρέπει να σταματήσουμε να σφίγγουμε τον πλοίο γύρω τους. Ένα άλλο θέμα Ξέρω ότι οι οικολόγοι και άλλοι στην Ευρώπη ε, επιθυμούν την συνέχιση της βιολογικής παραγωγής σε θερμοκήπιο. Είναι κρίμα ε, να μην βρεθεί λύση και να σταματήσει η σχετική παραγωγή. Επαναλαμβάνω, το, η ποιότητα του χώματος είναι θεμελιώδης σημασία και για μας. Θα πρέπει να μπορούμε να χρησιμοποιούμε χώμα που προέρχεται από πιο απόμακρες ε, περιοχές από ότι από όπου βρίσκεται ο παραγωγό. Αυτό το, η απέτηση του 80% για τοπικό χώμα είναι υπερβολική. Μόνο έτσι θα εξασφαλίσουμε την επιβίωση τη βιολογική παραγωγή και στι σκανδιναβικέ χώρε. Η κυρία Αγγιλέρα, ε, θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Χόισλινγκ το εξή. Όλα δείχνουν ότι πλησιάζουμε προ το τέλο των τριμερών διαλόγων. Αναφέρεται ότι 31 θα είναι ο τελευταίο τριμερής διάλογο. Αλλά παρόλα αυτά διαπιστώνω ότι έχουν παραμείνει πολύ σημαντικές διαφορές και εκκρεμότητες. Επειδή με η της γνωμοδότησης για τη Χιλή, ε, ζήτησα αναβολή της ψηφοφορίας της γνωμοδότησης, περιμένοντας την έκβαση των διαπραγματεύσεων για την επισήμαση των βιολογικών προϊόντων, ε, ελπίζοντας ότι θα ε, τελεσφορούσαν οι διαπραγματεύσεις. Είπατε ότι χρειάζεται καλή βούληση. Είναι, είναι πραγματικά πιθανό να καταλήξουμε σε κάποιο αποτέλεσμα σε αυτό το τελευταίο τριμερή διάλογο. Ε, γιατί εγώ δύσκολο το βλέπω. Και υπάρχουν κάποια καθόδη ζητήματα που, έχουν, που παραμένουν επίλυτα. Πιστεύετε πραγματικά πιθανό να ευοδοθεί ο τριμερής διάλογος στο εγγύς Είναι ρεαλιστικό να προσβλέπουμε σε διεκπαιρέωση και σε αίσιο πέρα στους ε, διαλόγους. Γιατί δεν αρκεί η αισιοδοξία, θα πρέπει να δούμε αν είναι ρεαλιστική αυτή η αισιοδοξία. Ευχαριστώ κύριε Νόιχλ. Ευχαριστώ. Μια συγκεκριμένη ερώτηση που την έχουμε συζητήσει για τα παραδοσιακά φάρμακα και ε, τις πρώτες ύλες για τα παραδοσιακά ε, αυτά προϊόντα συμπεριλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής ή όχι. Γιατί είναι σημαντικά, σημαντικό όταν ε, πάει στο φαρμακείο εφαρμογή ε, η οχι γιατι ειναι σημαντικο οταν παει στο φαρμακειο κανεις και αγορασει ενα τετοιο φαρμακο θα πρεπει να ξερει αν ειναι βιολογικη η παραγωγη εν προκειμένου θα είναι δηλαδή βιολογική παραγωγή αλλά δεν θα είναι η σήμανση βιολογική γιατί το ε, εμποδίζουν οι μεγάλες ε, ε, εταιρείες, οι φαρμακευτικές εταιρείες. Πιστεύω ότι πρέπει να λυθεί αυτό, ότι τα παραδοσιακά φυτικά φάρμακα θα πρέπει να έχουν οικολογική σήμανση όταν έχουν οικολογικά παραχθεί. Πώς έχει το θέμα τώρα. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Καλή τύχη εύχομαι για τον τελευταίο γύρο του τριμερούς διαλόγου. Όπως είπα και στην πρώτερη συζήτηση, δεν θα θρηνήσω αν τελικά καταρριφθεί αυτό το χαρτοφυλάκι. Προσπαθούμε να διορθώσουμε κάτι που δεν είναι σπασμένο. Αυτή η αγορά αυξάνεται σε όλη την Ευρώπη και βγάζουν χρήματα οι γεωργοί παράγοντας βιολογικά προϊόντα. Αυτό που δημιουργήσαμε είναι τεράστια βεβαιότητα. Έχουν σταματήσει οι επενδύσεις και το χειρότερο, προσθέσαμε και μαγικά στοιχεία στη συζήτηση. Πρώτα συζητήσαμε την αφαίρεση των κεράτων από τα, από το, τα ζώα, τα τροφία, που κάτι δεν είναι οικολογικό. Οικολογικό και βιολογικό σαν παραγωγή αφορά το να μην προσθέτεις ε, χημικά και να μην και να περιορίσει τη χρήση παρασετοχτών κλπ. Προσθέτουμε και κάτι μαγικό. Μετά το θέμα των εδαφών. Θα είναι να μην αγγίζουμε το χώμα. Θα είναι δύσκολο αυτό στο μέλλον αν έχουμε κάθετη γεωργία καλλιέργεια. Δεν θα γίνεται βιολογική αυτή η καλλιέργεια. Διότι στον 20ο όροφο δεν μπορεί να παράξει κάτι ε, χωρί να έχει ε, αγγίξει κανεί το χώμα. Τι είδου συζήτηση είναι αυτό. Ότι όλα πρέπει να προέρχονται από την ίδια εκμετάλλευση. Πάντα αυξάναμε την ποιότητα των εδαφών που χρησιμοποιούμε και οι γεωργοί πάντα ήταν πρακτικοί και ρεαλιστές. Αν έχεις πολύ καλό έδαφος και θες έχεις βιολογικό ο... υλικό, που αν το πετύψει καλό μηχάνημα, μπορώ ας πούμε να πάρω από σένα αυτό το χώμα, το βιολογικό υλικό που μας συντεθεί θα δημιουργήσει καλό χώμα και να το μεταφέρω στο δικό μου χτήμα. Όλα αυτά είναι ανοησία, ε, είναι κόλπα όλα αυτά. Δεν δημιουργείται μια ισχυρότερη αγορά για τα βιολογικά προϊόντα. Κάτι που ζητούν οι καταναλωτέ και θέλουν να πληρώσουν. Μιλάμε για περισσότερε επιδοτήσει για να παραχθούν προϊόντα από τη μια και από την άλλη θέλουμε να επιβάλλουμε περιορισμού σε πράγματα που λειτουργούν στην οικονομία τη αγορά με έναν τρόπο λογικό. Καλή τύχη σα εύχομαι. Αλλά όπω έθεσα και στο ερώτημά μου στον Επίτροπο, εγώ έθεσα μεγάλο προβληματισμό κυρίω για την ε, παραγωγή προκυπηστικών στι σκανδιναβικές χώρες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, πανέρχομαι στο θέμα των ε, πολυμάτων γιατί αυτό θα είναι η χειρότερη συμβαστική λύση μέχρι το 2022, μέχρι το 2025 θα υποβληθεί μελέτη, μετά δεν θα γίνει τίποτα για κάποια χρόνια, δηλαδή τα επόμενα δέκα χρόνια ε, δεν θα γίνει τίποτε. Οπότε, αν στην Ιταλία, για παράδειγμα, ένας ε, ε, βιολογικός καλλιεργητής ε, ε, κάνει, ε, παράγει σαλατικά και το, τα, τα υπολείμματα είναι πολλά, τότε δεν θα του αφαιρεθεί μόνο η άδεια, αλλά θα καταργηθεί και ε, το, το, το, προϊόν. Ε, σε μη βιολογικά μπορεί να είναι τα φυτοπροστατευτικά πενταπλάσια, αλλά ε, αυτήν την σαλάτα μπορεί να την ε, πουλήσει στις Ιταλικές αγορές. Οπότε τι γίνεται με την εσωτερική αγορά. Πιστεύω ότι είναι παράλογη η κατάσταση. Δεν είναι σωστοί οι κανόνες της εσωτερικής αγοράς ε, πώς το, το βιολογικό τομέας ε, αντιμετωπίζεται διαφορετικά εις ό,τι αφορά τα υπολείμματα. Ε, όταν δηλαδή ο καλλιεργητής βιολογικών έχει την ίδια ποσότητα ε, καταλήπων, ε, πώς ε, θα, ε, πώς θα αντιμετωπιστεί μετά ως καλλιεργητής βιολογικών προϊόντων. Το λέω αυτό γιατί ε, ε, το, το, θέμα αυτό δεν έχει αντιμετωπιστεί σωστά ούτε και από τις ενώσεις των καλλιεργικών βιολογικών προϊόντων. Νομίζω ότι εν προκειμένου η συμβιβαστική λύση που προτείνεται είναι παράδεκτη. Δεν έχουμε άλλους ομιλητές. Ο κύριος Χόισλινγκ πάλι. Ευχαριστώ συνάδελφοι και για τις παρατηρήσεις σας. Τώρα ε, αυτή η καταψήφιση είναι δύσκολη γιατί ξέρεις ότι η κατάσταση ε, είναι 50-50 σε ό,τι αφορά τα, τη βιολογική παραγωγή. Ε, υπάρχουν οριακές τιμές σε τρεις χώρες όπως είπα, διαφορετικές μάλιστα και οι περισσότερες ενώσεις δεν θέλουν οριακές τιμές καθόλου, ενώ στο Κοινοβούλιο η κατάσταση πάλι δεν είναι ξεκάθαρη, ε, για να το πω έτσι. Οπότε αυτό ε, δεν είναι υπεροπτική στάση. Αν η Κομισιόν ε, θέλει να θέσει κανόνες και αποφασίσουν οι περισσότεροι θα πρέπει να συμφωνήσουμε πάνω σε μια βάση. Η τελευταία συμβιβαστική λύση επί Προεδρίας ε, ήταν ένα κοκτέιλ τριών φυτοφαρμάκων και αν υπάρχουν τότε αφαιρείται η πιστοποίηση αυτομάτως. Τώρα, ποια βάση θα γίνει αυτό, πώς θα ε, γίνουν οι δειγματοληψίες, όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε. Επίση, το 50% ε, των ρήπων δεν έρχονται από την αγιοργία, αλλά από το εμπόριο, τη μεταποίηση και άλλους τομείς. Ε, ήδη υπάρχει ρήπανση αν χρησιμοποιήσουμε ένα φορτηγό για διαφορετικούς σκοπούς, τη μεταφορά διαφορετικών προϊόντων. Εμεί έχουμε ένα, στοιχείο, ένα κέντρο παρακολούθηση στη Βάδη Βιρτεμβέργη που είναι αποτελεσματικό και που δεν δείχνει μεγάλη επιβάρυνση, αλλά ε, δεν ε, χρησιμοποιούνται οι ίδιες μέθοδοι ε, σε όλε τις χώρες. Μπορεί όμως σε, για κάποια χρόνια να καλυφθούμε από αυτό, γιατί είναι χίλιοι ε, νομίζω ότι θα μετρήσει εδώ αν θα καταλήξουμε κάπου ή όχι, γιατί οι κανόνες για τις εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση σίγουρα θα γίνουν αυστηρότεροι. Συμφωνείτε ότι είναι σωστό για τον ευρωπαϊκό τομέα να τηρούν τους κανόνες μας και άλλοι, με ελάχιστε εξαιρέσεις βέβαια. Αλλά αυτό είναι και απέτηση των καταναλωτών, δηλαδή να υπάρχουν στα βιολογικά οι ίδιοι κανόνες και να τηρούνται από όλους. Ε, στο θέμα της θεματικής ε, παραγωγής ε, εδώ υπάρχουν κάποιες διαφορές υπάρχει δηλαδή ειδικό έδαφος για τη βιολογική καλλιέργεια κάποιοι επιμένουν σε αυτή την αρχή ε, έχουμε την οικολογική, βιολογική καλλιέργεια. Όταν αλλάξει η παραγωγή, ε, άμα την πούμε gardening για παράδειγμα και συνεχίσουμε, το, ε, μπορεί να αλλάξει η παραγωγή. Αλλά τότε δεν θα πρέπει η συνέχιση, ναι, αυτή η παραγωγή να χαρακτηρίζεται βιολογική ε, όταν θα παραμείνει στο έδαφος αυτό. Ε, δεν ξέρω. Ε, έχουμε εργαστεί πάρα πολύ σε αυτόν τον ε, τομέα και παρόλα αυτά ε, ενώ έχουμε έναν τομέα ο οποίος αυξάνεται και αναπτύσσεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θα έπρεπε κανονικά να υπάρχει μια εναρμόνιση στην αγορά. Ο τομέας αναπτύσσεται, αναπτύσσονται όμως και οι κίνδυνοι συμμετοχή στον τομέα αυτών ε, λάθος ανθρώπων. Γι' αυτό θα έπρεπε ίσως να υπάρχουν καμιά φορά πιο ενιαίοι κανόνες, ε, σε άλλες περιπτώσεις πιο αυστηροί, αλλά σίγουρα δεν θέλουμε να ε, καταπνίξουμε τον ε, αναπτυσσόμενο αυτό τομέα στην Ευρώπη. Α, συγγνώμη, αυτό είναι ένα από τα θέματα τα οποία συζητούνται και η συμβιβαστική λύση είναι καλή, αλλά είναι τα μικρά ανοιχτά θέματα που έχουμε και τα θα πρέπει να τα λύσουμε. Στο, στην ερώτηση που κάνατε, στο θέμα που θέξατε, μπορούμε να επανέλθουμε διμερώς. Ο κύριος Στάκουλα πάλι. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα παρακαλώ. Σε ό,τι αφορά για τις καλλιέργειες στο έδαφος, ε, Χθε όταν έφευγα από τη Φιλανδία χιόνιζε. Πώς να καλλιεργήσουμε στην Ήπεθρο, στο έδαφος. Με το ωραίο μας όμως θερμοκήπια καταφέρουμε να παράγουμε. Και είναι απαράδεκτο, μια και το χώμα που χρησιμοποιούμε στα θερμοκήπια μας είναι επίση από βιολογικές καλλιέργειε, να μην μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τα προϊόντα μας βιολογικά. Τι θέλετε, δεν εισάγουμε από τι Ηνωμένε Πολιτείε για να έχουμε μεγάλο αποτύπωμα περιβαλλοντικό αρνητικό. Αλλά το 80% που απαιτείται να είναι τοπικό χώμα είναι υπερβολικό. Στη Βιλανδία, ακόμη και στις κανονικές καλλιέργειες, ε, εδάφους, οι, οι δικές μας, οι συμβατικές καλλιέργειες είναι πολύ πιο καθαρές από τις βιολογικές καλλιέργειες της κεντρικής Ευρώπης, γιατί έχουμε πολύ λιγότερη μόλις του περιβάλλοντος, πολύ λιγότερη ατμοσφαιρική ρήπανση και ρήπανση του εδάφους. Ελπίζω πραγματικά ο κύριος Χόισλινγκ να μην οδηγήσει σε αφανισμό της βιολογικής γεωργίας στη Βόρεια Ευρώπη και ελπίζω στο μέλλον να μπορούμε να συνεχίσουμε και οι σκανδιναβικές χώρες να παράγουμε βιολογικά προϊόντα σε θερμοκήπια με καλό χώμα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χόισλινγκ και πάλι. Έχετε υποχρέωση τώρα να απαντήσετε, αλλά αν δεν το επιθυμείτε... Ε, δεν έχω πολλά να πω. Πήραμε και την επιστολή των πέντε υπουργών που θέλουν να ρυθμίσουν τις εξαιρέσεις. Είπα ε, ότι είτε θα διευρύνουμε τον κύκλο και θα είναι πιο περιοριστικές οι εξαιρέσεις ε, ή αν είναι ο 62ος παράλληλος τότε οι εξαιρέσεις δεν θα είναι ε, πολλές. Όταν πρόκειται για την αρκτική ζώνη, συμφωνώ μαζί σου, οι προϋποθέσεις είναι τελείως διαφορετικές. Αλλά για τη Σουηδία, για κομμάτια της Δανίας, δεν θα έλεγα ότι πρόκειται για περί αρκτικής ζώνης, οπότε γιατί θα πρέπει να υπάρξουν εξαιρέσεις από το γενικό κανόνα. Θα δούμε πού θα τραβήξουμε τη γραμμή. Πάντως θα λυθεί αυτό. Ε, βέβαια χρειάζεται και η σύμφωνη γνώμη των βορείων χωρών για μια συμβαστική λύση. Εύχομαι η αισιοδοξία σας ε, να μετατραπεί σε πραγματικότητα. Τι άλλο να πω. Η κατάσταση είναι δύσκολη. Και οι δικές μου ελπίδες είναι και δικές σας ελπίδες. Έχω κι εγώ, στις ελπίδες έχετε κι εσείς. Και νομίζω ότι αυτό αντικατοπτρίζει την πραγματική κατάσταση. Ότι έχουμε όλοι κοινέ ελπίδες. Τελευταίο θέμα, πολύ σύντομα, τρία λεπτά. 18 με 20 Απριλίου, ξέρετε, μετέβει η αποστολή μας στην Εστονία, προκειμένου να λάβουμε μέρος στο Αγροφόρου Μάρε Μπάλτικου και στην Διεθνή Γεωργική Έκθεση ΜΑΜΕΣ 2017 στο Τάρτου. Ε, η οργάνωση έγινε από την ε, γραμματεία της Επιτροπής ε, Άγκρη και τη μόνιμη αντιπροσωπεία της Εστονίας. Ξέρουμε περί τίνος πρόκειται, ήταν μέλη της αποστολής ο κύριος Μπόκοβιτς, ο κύριος Ντόρφμαν, ο κύριος Νέκοφ, η κυρία Μέλιορ, η κυρία Σένρα και ο υποφαινόμενος. Είναι η πέμπτη χρονιά που οργανώνεται το Αγκροφόρουμ, αυτή η Διεθνής Γεωρική Έκθεση. Πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση και σημαντική φωνή για τη γεωργία της περιοχής αυτής. Συμμετείχε μάλιστα και το Εστονικό Πανεπιστήμιο Βιοεπιστημών του Τάρτου. Συναντηθήκαμε με πολλούς ενδιαφερομένους και ε, υπουργού από τη Λιθουανία, τη Λετωνία, την Ουκρανία, τη Μολδαβία. Είχαμε πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και υπάρχει συνεργασία μεταξύ πολλών χωρών γύρω από τη Βαλτική και είναι πολύ αξιόλογες οι πρωτοβουλίες που γίνονται. Έχουμε πάρα πολλές γεωργικές εκθέσεις ε, ε, δασοκομείας, ε, γεωργίας, μεταποίησης πολιτών επαγγελματικού εξοπλισμού. Είχαμε γύρω στις 43.500 επισκέπτες και πάρα πολλά περίπτερα. Και χάρη στην αποστολή αυτή εξοικειωθήκαμε περισσότερο με την Γεωργία της Εστονίας και είδαμε τι αλλαγές έχουν γίνει. Μία στις τρεις ε, ε, α, α, είναι σε φάση εκαθάρισης. Αλλάζει το γεωργικό τοπίο στην Εστονία. Θα πρέπει λοιπόν ε, να δούμε και από αυτό το πρίσμα το μέλλον της κοινή πολιτικής. Ευχαριστούμε πάντως τη μόνιμη αντιπροσωπεία της Εστονίας και τη γραμματεία μας για την κοινή αυτή διοργάνωση. Θα σας στείλουμε τη σχετική τεκμηρίωση. Φαντάζομαι θα εξετάσετε με, το με πολύ ενδιαφέρον τα πορίσματα αυτής της επίσκεψης. Αυτά ολοκληρώνουμε αυτό το σημείο. Η επόμενη μας συνεδρίαση θα γίνει στις Βρυξέλλες 29 Μαΐου, 30 Μαΐου και 19 και 20 Ιουνίου. Επίση στις Βρυξέλλες. Αυτά, ολοκληρώνουμε. Τι να σου πω, καλό βράδυ. Σχεδόν φτάνουμε προς το τέλος της ημέρας. Καλή ξεκούραση πάντως. Γεια σας. Καληνύχτα.